I'm trying to sort of gently wait until there's one representative. Πρόεδρος, περιμένω μέχρι να έχουμε έναν εκπρόσωπο τουλάχιστον από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες. Ήλπιζα ότι θα βλέπαμε κάποιον από το ΕΛΚ που να ενδιαφέρεται για τους καταναλωτές και το πακέτο το σχετικό για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά δεν βλέπω. Βέβαια ξέρω ότι υπήρχαν πολλές συνεδριάσεις το μεσημέρι συγχρόνως. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Έχουμε βέβαια εδώ εκπροσώπους από σχεδόν όλες τις πολιτικές ομάδες, παρόλα αυτά. Και το επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι το πακέτο εκείνο το οποίο αποτελείται από την ανακοίνωση για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού διασυνοριακού εμπειρίου. Είναι πρόταση για τις υπηρεσίες παράδοσης των εμπορευμάτων βάσει του ηλεκτρονικού εμπορίου και είναι και το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού, αλλά και πρόταση κανονισμού όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών υπεύθυνων για τη συμμόρφωση όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Έχουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές για το δίκαιο εμπόριο, τις πρακτικές δηλαδή αυτές θέμη του εμπορίου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Τζέρατ Γκραφ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα περί του γεωγραφικού αποκλεισμού, έτσι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε για την ε, συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και στο τέλος θα ακούσουμε για την παράδοση των δεμάτων. Καλώς, ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους σας. Θα κάνω μία σύντομη εισαγωγή όσον αφορά τον γεωγραφικό αυτόν αποκλεισμό. Έχω κάτι διαφάνειες. Και αν εγώ στο τέλος ξεχάσω κάτι, τότε οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να τα συμπληρώσουν. Ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι βέβαια από μόνο του ένα σημαντικό μέτρο, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι είναι κομμάτι του πακέτου. Αν καταφέρουμε να, κάνουμε, να έχουμε μια πρόοδο είτε για την παράδοση των δεμάτων, είτε για την φορολόγηση, για το ΦΠΑ και θα κάνει σχετικά πρόταση η Επιτροπή μέσα στη χρονιά, τότε θα εξαφανιστούν πολλοί από τους λόγους για τους οποίους δεν καταφέρουν να πουλήσουν σε άλλες χώρες σε μέλη ή επιχειρήσεις μιας χώρας. Οπότε πρέπει να το δούμε το μέτρο και σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά και από μόνο του είναι σημαντικό. Και για ποιους λόγους. Θα μπορούσαμε να είχαμε το τριπλό παιχνίδι. Έχουμε το roaming που εξαφανίζεται από τον Ιούνιο, το θέμα της, μετα... της δυνατότητας μεταφοράς επίσης και του περιεχομένου προχωρούν και στο τέλος έχουμε και το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού. Αν αυτό προχωρήσει γρήγορα, αυτό θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όντως έχουμε τα εμπόδια και μπορούν πιο εύκολα να υποφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Το άλλο που θέλω να πω, γιατί έχουμε το θέμα το τι αιτιολογείται και τι δεν αιτιολογείται. Εδώ πέρα μιλάμε για γεωγραφικό αποκλεισμό που δεν έχει καμία αιτιολόγηση. Και ποια είναι η διαφορά, είναι ξεκάθαρη. Αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμό έχει να κάνει με περιπτώσεις που δεν πρόκειται για δυσκολίες που έχουν οι έμποροι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή τα αγαθά τους σε πολίτες που κατοικούν σε άλλη χώρα. Αν είναι πιο περίπλοκο, όπως συμβαίνει αν πρέπει να ε, μεταφέρει το εμπόρευμα σε μια άλλη χώρα ο έμπορος, ε, τότε εντάξει, υπάρχουν και έξοδα, τότε μπορούμε να πούμε ότι αιτιολογείται. Αλλά ελπίζουμε ότι με τα άλλα μέτρα τα οποία προωθούνται, τότε ό,τι λόγοι παραμένουν που δικαιολογούν κατά κάποιο τρόπο τις δυσκολίες, δεν θα έχουμε πια. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου είναι τελώς αδικαιολόγητο και αυτό ακριβώς είναι που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ. Περιλαμβάνονται όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Γιατί εκεί ακριβώς είναι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει μέτρα για να διευκολύνει την προσφορά υπηρεσιών. Είναι πιο εύκολο δηλαδή σε διασυνορικό επίπεδο να προσφέρονται υπηρεσίες. Τώρα, ποιες υπηρεσίες δεν καλύπτονται αυτές που δεν καλύπτονται από την υπηρεσία, για τις, από την οδηγία για τις υπηρεσίες, τα οπτικοακουστικά. Αυτά τα εξετάσουμε σε ένα διαφορετικό κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπό το copyright. Οι υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικά, έχουν τη δικιά τους λογική, οι μεταφοράς, εκεί οι αρχές είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, εκτός από τους σιδηροδρόμους δηλαδή, κομμάτι του κοινοτικού κεκτημένου. Τηλεπικοινωνίες, ούτε αυτές καλύπτονται. Οι αδικαιολόγητες περιπτώσεις τώρα γεωγραφικού αποκλεισμού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει πολλή δουλειά με διαβουλεύσεις, με μελέτες, για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Μιλάμε για καταστάσεις όπου οι έμποροι επίτηδε προσπαθούν να κατακαιρματίσουν την αγορά. Και από την μελέτη που κάνουμε, όντως υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, πάνω από 10.000 ε, ιστοσελίδες. Και φαίνεται ότι 8 με 30% όλων των συναλλαγών ε, των ηλεκτρονικών εμπορικών τελικά εμποδίζονται, δηλαδή δεν καταλήγουν επειδή υπάρχει μια προσπάθεια από τους εμπόρους να κατακαιρματίσουν την αγορά. 75% πρόκειται για δικαιολογημένους λόγους, γιατί όντως χρειάζεται κάτι παραπάνω, αλλά σε 25% των περιπτώσεων επίτηδες οι έμποροι δεν εξυπηρετούν ένα πολίτη που βρίσκεται σε άλλη χώρα, γιατί οικονομικά τους συμφέρει να κατακαιρματίζουν την αγορά. Έχουμε εντοπίσει πέντε περιπτώσεις που πιστεύουμε ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός δεν δικαιολογείται, τέλος πάντων δεν δικαιολογείται πια. Το ένα είναι ο αποκλεισμό ή το rerouting που γίνεται ώστε να καταλήξει στην ιστοσελίδα μιας άλλης χώρας ε, μέλους. 2% των ιστοσελίδων που είναι 8% του, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Δηλαδή τι λέμε εδώ, λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιος αποκλεισμό εκτός αν υπάρχει κάποια εθνική ρύθμιση που απαιτεί τον αποκλεισμό αυτό. Και δεν πρέπει αυτόματα να οδηγήσει τον πελάτη αλλού. Πρέπει να συμφωνήσει ότι θέλει να μεταφερθεί στη δικιά του τη χώρα ή κάπου αλλού. Η δεύτερη περίπτωση είναι όπου κάτι που βλέπεις πολύ καλά και στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή πας σε ένα κατάστημα σε μια άλλη χώρα, κανένας δεν θα σε ρωτήσει από πού προέρχεσαι και θα σου πει δεν θα σε εξυπηρετήσω επειδή είσαι από μια άλλη χώρα. Αν λοιπόν ένα πελάτη θέλει να κάνει μια παραγγελία σε άλλη χώρα, επιθυμεί να τύχει τη ίδια μεταχείριση σαν να ήταν κάτοικος τη άλλη χώρα. Οπότε να μπορεί να πάρει το πράγμα που παράγγειλε ο πελάτης χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα έπρεπε λοιπόν να μην υπάρχει ούτε και εδώ ο γεωγραφικός αυτός αποκλεισμός. Η τρίτη περίπτωση είναι όταν διασυνοριακά πρέπει να ε, παραδοθούν υπηρεσίες. Cloud είναι πολύ πιο εύκολο να προσφέρονται online υπηρεσίες από ότι σε φυσική μορφή. Λέμε ότι δεν είναι κάτι περίπλοκο. Οι υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να διατίθεται ε, εφόσον το ζητάει ο καταναλωτής στη χώρα του. Έχουμε βέβαια προβλέψει κάποιες εξαιρέσεις γιατί πρέπει να εφαρμοστεί το ΦΠΑ της χώρας του πελάτη. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια νομική περιπλοκότητα ακόμα. Η τέταρτη περίπτωση είναι κάτι που έχουμε ακούσει και το έχουμε ίσως και ζήσει, όπου η ίδια υπηρεσία όταν καταναλώνεται κατά από τις ίδιες συνθήκες ε, στο χώρο που βρίσκεται ο πελάτης, ε, πληρώνεται σε διαφορετική τιμή από, όταν, ε, από όπου κατοικεί ο καταναλωτής, από όπου το παραγγέλνει, είτε πρόκειται σε ένα ξενοδοχείο, είτε κάπου αλλού. Πιστεύουμε ότι και αυτό είναι κάτι αδικαιολόγητο. Και αυτό ισχύει για όλα, ότι οι τιμέ, έτσι κι πρέπει να είναι ίδιε σε όλε τι χώρε μέλη. Οι επιχειρήσει μπορεί να έχουν ιστοσελίδε με διαφορετικέ τιμέ σε μία χώρα μέλο, έχει νόημα, αλλά αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσει, είναι όταν θέλουν οι καταναλωτέ να αποφεληθούν από μία ευνοϊκή τιμή σε άλλη χώρα, να υπάρχει αυτός ο γεωγραφικός αποκλεισμός και να μην μπορούν να έχουν αυτή την ευνοϊκή τιμή δεν μπορείτε να εμποδίζετε τους καταναλωτές να υποφεληθούν από μια πιο ευνοϊκή τιμή επειδή ζουν σε μια διαφορετική χώρα. Τέλος υπάρχει για το θέμα του τρόπου πληρωμής. Από την δικιά μας ανάλυση σε πολλές περιπτώσεις περνάτε από όλη τη διαδικασία για την παραγγελία και τελικά δεν γίνεται δεκτός ο τρόπος πληρωμής που διαθέτεις. Τον απορρίπτει το σύστημα. Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος οι έμποροι να αρνούνται μέσα πληρωμής τα οποία δέχονται από τους κατοίκους της χώρας όπου είναι οι εγκατεστημένοι, αλλά δεν τα δέχονται από κάποιον που πληρώνει από μια διαφορετική χώρα. Αυτές είναι οι πέντε περιπτώσεις. Θα ζητήσω από τον Γιούργεν να εξηγήσει λιγάκι τι σχέση έχουν όλα αυτά με την οδηγία για τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές του νόμου, γιατί με αυτά θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, ναι, το σημείο κίνησης είναι γιατί χρειαζόμαστε αυτό τον κανονισμό. Έχουμε ήδη το άρθρο 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Είναι θέμα αρχής μη διάκρισης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις, αλλά στην πράξη τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό δεν το γνωρίζαμε. Το 2012 προσπαθήσαμε να πιέσουμε τις χώρες μέλη να αναλάβουν δράση. Δεν έγινε τίποτα. Είχαμε πολλές προσφυγές. Συνεπώς είναι σημαντικό ότι δεν θα τροποποιήσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες, γιατί είναι ένα λέξ σπεσιάλης, όπως το λέμε, ένα ειδικό νομικό μέσο, το οποίο ισχύει και προσφέρει και την απαραίτητη νομική σαφήνεια σε περιπτώσεις όπου πιστεύουμε ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός δεν δικαιολογείται. Δεύτερη παρατήρηση. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και με τους εμπόρους. Αν έρθει σε επαφή μαζί μου ένας καταναλωτής από μια άλλη χώρα και κληθώ να παραδώσω ένα προϊόν, βάσει των όσων σας περιγράψαμε πριν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δω τι ισχύει, τι εφαρμόζεται ως νόμος για τους ξένους. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Εμείς ε, τη Ρώμη 1, τη συμφωνία αυτή, δεν την αγγίζουμε. Θέλουμε νομική ασφάλεια. Αν είσαι μια μικρομεσαία επιχείρηση, σε μια μεγάλη χώρα μέλος, δεν επηρεάζεσαι από την ομοθεσία για τους ε, ξένους και ελπίζουμε έτσι κι αλλιώς να υπάρξει σύντομα ευρωπαϊκός νόμος. Η διάταξη 1 του μέσου αυτού είναι πολύ σημαντική για τους εμπόρους, γιατί τους προσφέρει νομική ασφάλεια. Εμείς δεν θέλουμε να μειώσουμε την προστασία του καταναλωτή. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να διευκρινίσουμε πού ακριβώς βρίσκεται ο έμπορος μέσα σε όλα αυτά τα νομικά μέσα. Βέβαια μετά έχουμε να κάνουμε και με την παράδοση των αγαθών. Η συνάδελφος από την προστασία καταναλωτών όμως θα σας μιλήσει γι' αυτά. Ευχαριστώ. Θα μας μιλήσετε για τον κανονισμό όσον αφορά τη συνεργασία για την προστασία καταναλωτών, σωστά? για να συμπληρώσουμε αυτό το πακέτο συμπεριλάβαμε πω είχε προαναγγελθεί για τη στρατηγική τη ενιαίας αγορά, την αναθεώρηση για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία καταναλωτών υφιστάμενο από το 2004 μέσο και έχει τον μοναδικό ε, χωριστό χαρακτήρα για την νομοθεσία για την ενιαία αγορά που επιβάλλει συνεργασία μεταξύ των αρχών ώστε να επιβληθούν μέτρα στα διασυνοριακά θέματα σε 30 ε, θεματολογικά ζητήματα, ξεκινώντας όσον αφορά τις πρακτικές συμβάσεις ε, και όρους ε, συμβάσεων, τα δικαιώματα καταναλωτών κτλ. Ήταν ένας κανονισμός αυτός, μια ρύθμιση, αλλάζει η διαφάνεια. Μια στιγμή πήγε πολύ γρήγορα. Ζήτω συγγνώμη γι' αυτό. Οι ρυθμίσεις από το 2004 ισχύων Για τη διασυνοριακή παραδοσιακή συνεργασία χρησιμοποιήθηκε, αλλά όχι στο μέτρο του πλήρους δυναμικού. Και θεωρήσαμε ότι ήρθε επιτέλους τώρα η χρονική στιγμή να αναθεωρήσουμε αυτή την νομοθετική πρακτική, αυτό το πλαίσιο, να δούμε τις ελάχιστες δικαιοδοσίες και εξουσίες που έχουν τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να αυξηθεί το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους Πρέπει επίση να επεκταθεί το εύρο, το φάσμα, ώστε να ενταχθούν και περισσότερα θέματα νομοθετικά. Καθώς επίσης και η πρόταση για την ε, κατάργηση των γεωγραφικών αποκλεισμών. Θέματα που δεν εντασσόντουσαν σε αυτό το φάσμα. Και πώ θα συντονιστούμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ευρύ φάσμα παραβάσεων και παραβιάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι μέχρι σήμερα έχουμε ισχυρές οργανώσεις και συλλόγους καταναλωτών, αλλά δεν συμβαίνει αυτό σε όλα τα 28 κράτη-μέλη. Μάλιστα μόνο σε μια μειοψηφία, μειονότητα κρατών μελών ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν διέπουν την πρότασή μας για μια αναθεώρηση, επανεξέταση. Τι πετύχαμε μέχρι σήμερα με τον ενισχύ κανονισμό. Θα θυμόσαστε την περιβόητη περίπτωση κατά των μεγάλων πλατφόρμων. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η διαφάνεια για την κατάργηση της αγοράς ε, δωρεάν όσον αφορά τα παιχνίδια για τα παιδιά, ενώ έπρεπε να γίνονται κάποιες αγορές. Καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο χρησιμοποιώντας την, ε, το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις, όπου καταφέραμε να πείσουμε και την Amazon και την Google και την Apple να άρουν, να απαλείψουν τον όρο free δωρεάν από αυτές τις προσφορές τους εν ώψη και της οδηγίας ε, για τα δικαιώματα ε, των καταναλωτών. Καταφέραμε επίσης να πείσουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες να αλλάξουν τους όρους και προϋποθέσεις και να ε, τους ζητήσαμε να επανέλθουν στις ε, ε, πρακτικές ε, για τις οποίες δεν γνώριζαν οι καταναλωτές αλλά αποκαταστάθηκε το καθεστώς που επιθυμούσαμε. Αυτό ήταν αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. Επίσης και το SWEEP η εξέταση, ο έλεγχος εκατοντάδων ιστοσελίδων. Καταφέραμε να διορθώσουμε πάρα πολλές τέτοιες ιστοσελίδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και κατάρτιση, εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών που είναι σημαντικός όρος και προϋπόθεση για το ισοδίκαιο πλαίσιο εφαρμογής, level playing field. Γιατί πρέπει όλα αυτά να γίνουν. Σε μια μελέτη που έγινε εξέταση για τις μελέτες επιπτώσεων είδαμε ότι 37% του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ε, ε, ιστοσελίδων δεν σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών υπό το 5E. E. Κάναμε αυτή την επισκόπηση ένα 1Ε Electronics. Δεν γνωρίζω γιατί σε τι οφείλεται ότι δεν μπορεί να παρουσιαστεί η διαφάνεια. Εν πάση περιπτώσει. λοιπόν του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ε, συμβάσεων δεν σέβονται τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών για τα ε, ρούχα, τον ηματισμό, ε, χρηματοοικονομικά, ε, ηλεκτρονικά. Υπάρχουν σημαντικοί τομείς όπου δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των καταναλωτών και πρέπει να αντιμετωπιστούν τέτοιες παραβιάσεις και παραβάσεις. Υπολογίσαμε κάτι τίμηση 770 εκατομμύρια είναι, τα είναι το ποσό που ζημιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να μπορούν να είναι σεβαστά αυτά από τους συναλλασσόμενους. Τώρα, πώς θα αλλάξουν αυτά και πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα με τη νέα πρόταση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σήμερα οι αρχές, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ γιατί δεν αλλάζει η διαφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Λοιπόν, στην οθόνη πάλι. Σήμερα οι αρχές μπορούν να αντιδράσουν μόνο κατά των αυξανόμενων παράνομων πρακτικών. Αν υπάρχει μια ιστοσελίδα που σας προσέφερε κάτι, αλλά δεν υπάρχει πια αυτή η προσφορά. Δεν μπορούμε αναδρομικά να ασκήσουμε δίωξη σε σχέση με, την, ε, ε, με, κάτι το παραπλανητικό. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτή η συνιστός ότι αναδρομικά αν έχει κάτι αλλάξει δεν μπορεί να διωχθεί. Για κάποιους άλλους τομείς όπως αναφέραμε το φάσμα της νομοθεσίας που κάλυπτε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ε, νομικές, αλλά όχι και την, τον γεωγραφικό αποκλεισμό και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και το άρθρο 20 της Οδηγίας περί Έχουν περιορισμένες εξουσίες οι αρχές ε, για να ε, δράσουν. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να προσπαθήσουμε να δράσουμε, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, οι αρχές να δράσουν διαφορετικά εναντί των συναλλασσόμενων, στο πλαίσιο του εμπορίου ώστε να υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες σε σχέση με τους ιδιοκτήτες αυτών των ιστοτόπων και να υπάρξει πλήρης αποζημίωση για την οποιαδήποτε ζημιά. Πιο σημαντικό να αντιμετωπιστούν ευρύτατες πρακτικές που δεν αντιμετωπίζονται συντονισμένα και ενιαία σήμερα. Εισάγουμε στη διαδικασία ένα νέο επίπεδο ενιαίας μορφής που θα ε, βρίσκεται υπό, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον διαθρωμένο δομημένο διάλογο έγινε λόγος για τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται με αυστηρό τρόπο για αυτές τις διεργασίες. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για την αντιμετώπιση των παραβάσεων και παραβιάσεων στην Ευρώπη. Και τελευταίο εξίσου σημαντικό για τις ενώσεις και συλλόγους για τα δικαιώματα των καταναλωτών θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα από πλευρά τους να δράσουν και να δίνεται μια έγκαιρη προειδοποίηση. Κάποια παραδείγματα που έχουμε δώσει σε αυτή τη διαφάνεια, αλλά που δεν φάνηκε έγκαιρα, για παράδειγμα, για κάποιες προσφορές στον τομέα των ε, ε, αεροπορικών μεταφορών με πακέτα όπου υπάρχει για παράδειγμα μια ε, περιορισμένη προσφορά λίγων ημερών αλλά όταν διαπιστώνει κανείς ότι η τιμή έχει αλλάξει επειδή δεν ισχύει πλέον όπως εκείνη την ημέρα προσφοράς έναντι τέτοιων πρακτικών θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Και για συνδρομές ε, που έχει ε, συμβατικά συνάψει κάποιος χωρίς να γνωρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει, τώρα όλες αυτές οι περιπτώσεις θα καλύπτονται από την ομοθεσία. Το υλικό το οποίο διαχέεται από το ένα κράτος στο άλλο, πράγμα το οποίο θα πρέπει σε ένα ενιαίο πλαίσιο να μπορεί να γίνει, θα μπορούμε να το πετύχουμε. Πανενοσιακά λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και προσφυγές ε, για την μίσθωση αυτοκινήτων για παράδειγμα, 8.000 τέτοια παράπονα που είχαν κατατεθεί και πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο να μπορούμε να δράσουμε. Ένα παράδειγμα για, για αυτή την ε, ε, ευρύτερη περίπτωση παραβιάσεων, μια γνωστή εταιρεία, αντί για την ελάχιστη περίοδο δύο ετών εγγύησης που <clears throat> θα είχε δικαίωμα να διεκδικήσει ο καταναλωτής καλύπτει για ένα έτος το προϊόν και μπορεί να αγοράσει την επέκταση της εγγύησης για άλλο ένα έτος ο, ο καταναλωτής. Απαράδεκτο αυτό. Αν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη νέα διαδικασία ως Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταχρηστικές πρακτικές. Ποια είναι τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και ωφέλη για τους καταναλωτές εν κατακλείδη. Υπάρχει για παράδειγμα αντιστάθμιση, αποζημίωση. Θα σταματήσουν ταχύτερα τέτοιου είδους πρακτικές. Θα υπάρξει κύρωση για τέτοιου είδους πράξεις ε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τις επιχειρήσεις θα ε, πάψει να υπάρχει ε, σημαντικός ε, ρόλος κάποιων εταιριών και θα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θα μπορούν να συνεργαστούν ισχυροί παίκτες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Υπολογίσαμε 45% του κόστου συνολικά μπορεί να εξοικονομηθεί μέσω συντονισμένων δράσεων καθώς επίσης και λόγω της εξοικονόμησης του κόστους διατησίας που δεν θα χρειαστεί να επακολουθήσει, όπως είπα μέσα σε ένα πλαίσιο level playing field, ενός ισοδίκαιου πλαισίου δράσης και δραστηριοποίησης. Και για αυτό το τμήμα του, της δέσμης μέτρων για την επιβολή μέτρων και τις κυρώσεις δεν μπορώ να τονίσω επαρκώς τη σπουδαιότητα αυτού του ε, μέτρου. Είναι ακριβώς ο ακρογωνιαίος λήθος και έχει πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν κάλυπτε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Γνωρίζουμε από συλλογή στοιχείων ότι 44% των καταναλωτών λένε ότι συνάντησαν παραπλανητικές τέτοιες περιπτώσεις σε διαφημίσεις ε, ή σε προσφορές ε, κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Σχεδόν 25% λένε ότι αγόρασαν κιόλα ένα τέτοιο προϊόν. Πραγματικά είναι πρόβλημα αυτή η κατάσταση. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο και την πείρα που συλλέξαμε υπό το CPC η περίπτωση, η περίπτωση που αφορά τις ε, μη θεμητές πρακτικές στο εμπόριο. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο και γι' αυτό καταλήξαμε με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ε, και κατευθύνσεις ε, που θα γνωρίζουν ακριβώς οι εταιρείε Ποιο είναι ο νόμος και πώς πρέπει να εφαρμόζεται. Οι αρχές ε, ε, και οι σύλλογοι ενώσεις για την προστασία καταναλωτών θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν ώστε να εφαρμοστούν όλες αυτές οι αρχές. Δύο πολύ ζωντανά παραδείγματα που θα ήθελα να σας αναφέρω. Για παράδειγμα, τι λέγεται σε σχέση, τι γίνεται σε σχέση με εκείνους που ως ε, συναλλασσόμενοι συμμετέχουν στο εμπόριο. Είναι συνεισφορά μας στο εμπόριο αυτό για να γνωρίζουν όλοι τι συμβαίνει με τη δραστηριοποίηση εμπλεκόμενων σε πλατφόρμες. Και έχουμε ένα τέτοιο καλό παράδειγμα. Για παράδειγμα από την Ιταλική Αρχή για τον Ανταγωνισμό, απόφαση του 2014, όπου η Αρχή για τον Ανταγωνισμό και την Προστασία Καταναλωτών είπε ηλεκτρονικό εμπόριο ενός διαμεσολαβητή που παρήχε υπηρεσίες ηλεκτρονικά ήταν, ένας, ε, ήταν μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν περιοριζόταν σε ε, απλή ενημέρωση αλλά σε προσφορές, σε ε, εστιατόρια, ακόμα και την δυνατότητα σε εισαγωγικά συγκρίσεων όπως αναφερόταν. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό τμήμα κατευθυντήριων γραμμών αυτό. Ένα άλλο παραπλανητικές δηλώσεις ε, για την περιορισμένη ισχύ ή ε, τις ιδιότητες ενός προϊόντος όταν αγοράζετε ένα εισιτήριο, όταν ε, κλείνετε δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, όταν υπάρχουν απουσίες ή ελλείψεις από πλευράς εισιτηρίων ή κρατήσεων, μπορεί να είναι όλα αυτά παραπλανητικά και να αποβαίνουν προς εις βάρος ε, των καταναλωτών. Και γι' αυτό αποφασίστηκε ότι η, μη ενημέρωση των καταναλωτών για τα διαθέσιμα προϊόντα μπορεί να αποτελεί παραπλάνηση. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στο στον ηλεκτρονικό ψηφιακό κόσμο. Δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία, νέες κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει μέσα στο πλαίσιο αυτό των υφιστάμενων να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. And on parcel delivery from Furnace Καλησπέρα σε όλους. Περιμένω ακόμα τις διαφάνειες. Οπότε η διασυνοριακή αποστολή δεμάτων και ο αντίστοιχο κανονισμός δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν προετοιμαστήκε στα γρήγορα. Έχει πενταετή ιστορία και η παρουσά επιτροπή ενεπλάκη σε όλες τις προπαρασκευαστικές φάσεις από τότε που το 2012 εντοπίσαμε τα βασικά ζητήματα. Η αποστολή δεμάτων έγινε ένα κεντρικό ζήτημα τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Προχωρήσαμε το 2012 στην Πράσινη Βίβλο, η οποία επιβεβαίωσε πως αποτελεί πρόβλημα. Αλλά υπήρξαν έντονα σήματα από τις αγορές, από το Κοινοβούλιο, από τα κράτη-μέλη, πως θα έπρεπε να βασιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην αγορά και όχι να ρυθμίσουμε γρήγορα. Ένα χρόνο αργότερα είχαμε τον οδικό χάρτη, στον οποίο εντοπίσαμε ζητήματα όλων των ειδών, από την οπτική γωνία της αποστολής, η τιμή, η διαλειτουργικότητα και άλλα. Το κάναμε με ένα πνεύμα συνεργασίας, καλέσαμε τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως και τα κράτη-μέλη, να θεσπίσουν μέτρα, να προσκομίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό που έχετε τώρα μπροστά σας είναι ένα σχέδιο κανονισμού που προσπαθεί να επιδιορθώσει κάποια τμήματα από τον αρχικό ορισμό του προβλήματος που δεν αντιμετωπίστηκαν από κάποια άλλα μέτρα που ελήφθησαν. Έχουμε κάποια παραδείγματα στη διαφάνεια εδώ όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα παραδείγματο χάρη. Έχουμε έντονες επενδύσεις στην βελτίωση της συνεργασίας εάν χρησιμοποιεί κανείς δύο μεταφορής, για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την αγορά. Παρακολουθούμε από στενά τι γίνεται. Οι λιανοπολιτές επίσης συμπεριέλαβαν νέα ζητήματα στα σήματα εμπιστοσύνης τους. Επίσης συγχρηματοδοτήσαμε το τελευταίο σημείο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ενημέρωσης μέσω του κόσμου. Ήταν το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βλέπουμε λοιπόν πως συμβαίνουν πολλά, τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως δεν θα πρέπει να δράσουμε τώρα. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν μείωσε το πρόβλημα που πάντα ξεχώριζε σε οποιαδήποτε διαβούλευση με καταναλωτές ή επιχειρηματίες, που είναι το κόστος των διασυνοριακών αποστολών. Στη διαφάνεια βλέπουμε παραδείγματα. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό πολιτών και αγοραστών όταν τους ρωτήσει κανείς. Αναφέρουν το κόστος, την τιμή της αποστολής αλλά και της επιστροφής αγαθών ως πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να βελτιώνεται καθώς περνάει ο χρόνος. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πρόταση τώρα προδιαβούλευση στο τραπέζι σας. Η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας αυτής, και αυτό είναι σημαντικό, είναι πως πιστεύουμε ακόμα πως οι δυναμές της αγοράς είναι οι καλύτερες για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Είναι ένα συνοδευτικό μέτρο το οποίο συνοδεύει όλες τις λύσεις που βασίζονται στην αγορά που προανέφερα. Είναι ένα πολύ στοχευμένο μέτρο που εστιάζει αποκλειστικά στην τιμή, στην ρυθμιστική εποπτεία και στην πρόσβαση, που σημαίνει μια βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς. Επίσης ενισχύει τη θέση των ευάλωτων καταναλωτών ή μάλλον μικροπολιτών και όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά για πολύ μικρές επιχειρήσεις ή για πολίτες τους οποίους δεν προσφέρονται προσιτές τιμές διασυνοριακά. Και τρίτον, επίσης λάβαμε, το θεωρήσαμε ως ένα πολύ ισορροπημένο μέτρο. Δεν θα έχουμε ρύθμιση τιμών. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μέσω της διαφάνειας. Είτε για τους πολίτες, είτε για τους ρυθμιστές. Δεύτερον, προσπαθούμε να διατηρήσουμε το διαχειριστικό φράγμα στο ελάχιστο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για την εκτέλεση του κανονισμού αυτού. Όπως βλέπετε από την δομή του κανονισμού, βλέπετε ότι θα είναι πολύ λεπτός. Είναι μόνο κάποια λίγα άρθρα. Παροχή πληροφοριών, άρθρο 3, μετά το άρθρο 4, 5, 6, ασχολούνται περισσότερο με τις επιχειρήσεις, στο άρθρο 9 επίσης βλέπουμε λίγη επιτροπολογία. Εκεί προσπαθούμε να, να διασφαλίσουμε πως τα αιτήματα ενημέρωσης που θα απευθύνονται στις επιχειρήσεις θα είναι τα αναγκαία, αναλογικά, αλλά επίσης όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένα. Επειδή εάν είστε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον πανευρωπαϊκό τομέα της εφοδιαστικής, κάτι διαφορετικό δεν θα προωθούσε το αντικείμενο της δραστηριότητάς σας. Το άρθρο 3 θα δίνει την εξουσία στους ρυθμιστές να κοιτάξουν όλη την αγορά και όχι μόνο την κλασική ταχυδρομική αγορά. Εάν ρίξετε μία ματιά στις αγορές αυτές, θα δείτε ότι όντως υπάρχει πολλής ανταγωνισμός. Πολλά διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που είναι δύσκολο να συγκριθούν το ένα με το άλλο. Έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, integrators, που παραδοσιακά ε, παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αν και είναι ακριβές. Και έχουν πολλές διαφορετικές τιμές, δομές τιμολόγησης, έχουμε τις εθνικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, έχουμε πανευρωπαϊκά δίκτυα αποστολής, που συχνά αποτελούνται από εθνικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις, έχουμε εγχώριους μεταφορείς, αλλά επίσης περισσότερους παράγοντες που μπαίνουν όπως μεγάλοι πολιτές της Λιανικής, που μπαίνουν επίσης στον χώρο αυτό. Ωστόσο, οι ρυθμιστές μας παραδοσιακά είχαν μόνο την εξουσιοδότηση, την εξουσία, να κοιτάξουν τις εθνικές αγορές και οι ρυθμιστές μας είπαν επανειλημμένα πως υπάρχουν προβλήματα νομικής σαφήνειας, βεβαιότητας έλλειψης δεδομένων, έλλειψης εξουσιών, για να μπορέσουν να εντοπίσουν ζητήματα ανησυχίας σε αυτή την αγορά που αλλάζει τόσο γρήγορα. Αυτό είναι λίγο η λογική πίσω από την πρόταση αυτή. Πιστεύω πως εύκολα μπορούμε να αποδείξουμε πως η αποστολή είναι κρίσιμη σημασία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Χαρακτηρίζεται από το νόγκο τη, το οποίο σημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρχουν ατέλειωτοι αριθμοί επιχειρήσεων εκεί έξω. Δηλαδή η ισχύ της αγοράς θα επηρεάσει την εμπορική δραστηριότητα. θα πρέπει να αρχίσουμε χρησιμοποιώντα άλλα τμήματα των δικτύων. Έχουμε αγορέ που αλλάζουν γρήγορα, που μετακινούνται γρήγορα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα με διαφορετικέ νομικέ απαιτήσει και διαφορετικά υπόβαθρα. Το ζήτημα των ίσων συνθήκων για όλους αποτελεί ένα πρόβλημα όσον αφορά την συμπεριφορά κάποιων από αυτές τις επιχειρήσεις. Όταν περάσουμε στο ζήτημα της προσιτότητας, το ζήτημα αυτό αφορά αποκλειστικά τους ευάλωτους καταναλωτές και όχι όπως είπα πριν όλες αυτές τις, ε, αυτά τα διαπραγματευμένα τιμολόγια, κοστολόγια. συνήθως πρόκειται για επιχειρηματικά μυστικά ή τα συνήθη κοστολόγια, τα οποία συνήθω δεν αποτελούν πρόβλημα. Αλλά εάν είστε πολίτης ή μικρός λιανοπολιτής δεν έχετε επιλογή. Ακόμη και αν υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις, αυτές τείνουν να εστιάζουν στους, στις μεγάλες επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά όχι στους μικρούς λιανοπολιτές, ιδίως όχι στην περιφέρεια. Και έτσι οι πολίτες βασίζονται κυρίως στις εθνικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Και εκεί οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Έχουμε πολλές ενδείξεις για στρέβλωση των τιμών. Δεν μπορείτε να το δείτε από εκεί, εγώ μπορώ. Το μήνυμα είναι όμως πως οι διασυνοριακές τιμές είναι κάποιες φορές κατανοητά υψηλές. Είναι τρεις έως πέντε φορές υψηλότερες από τις εθνικές, τις εγχώριες. Βλέπω ότι η ταχυδρομική υπηρεσία αφαίρεσε τη διαφάνειά μου. Συχνά δεν υπάρχουν σαφείς λόγοι για το κόστος αυτό και θα συνεχίσω χωρίς τη διαφάνεια. Έχουμε πολλές μελέτες που αποδεικνύουν. Συγγνώμη μια στιγμή. Διατίθεται ακόμα από την εφαρμογή e-meeting στο λάπτοπ σας ή στο τηλέφωνό σας. και πιστεύω πως, πως μπορείτε να μπείτε άμεσα μέσω το Q-Card στο, στην εφαρμογή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εντυπωσιασμένο από τι διαδικτυακέ ικανότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο η παρούσα επιτροπή, καμία άλλη. Φυσικά, φυσικά. Λιγότερο εντυπωσιακέ είναι οι τιμέ των διασυνοριακών δεμάτων, που είναι 3 5 φορές υψηλότερες από τις εγχώριε, κάποιες φορέ αυτό είναι κατανοητό. Αν συγκρίνει κανεί αποστολέ από το Βέλγιο, από τι κάτω χώρες, οι τιμές των κάτω χωρών είναι οι διπλασιέ από του Βελγίου. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδειγμάτα. Υπάρχουν μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Σαντ Λούις, που ασχολούνται με το υψηλό επίπεδο τιμών αλλά και την απουσία αιτιολόγησης για το κόστος αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Εάν δηλαδή αυτό οφείλεται στη μεταφορά ή σε οτιδήποτε θα εξηγούσε τις τεράστιες αυτές διαφορές. Εάν πρόκειται δηλαδή για έλλειψη ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο μερίδιο της αγοράς. Η κατανόηση της δομής του κόστους Μα δείχνει πως το κόστος μεταφοράς αναδέμα είναι περιορισμένο. Το τελευταίο τμήμα ασχολείται με την πρόσβαση, όπως είπα προηγουμένως. Εάν αρχίσετε να μπαίνετε σε νέε αγορέ, τότε θα χρησιμοποιήσετε υφιστάμενα δίκτυα. Και εδώ θα σπίσαμε νέε υποχρεώσεις. Επικοδομούμε σε αυτό που είναι έτοιμο, αλλά δεν λειτουργεί, γι' αυτό και προσπαθούμε να επισκευάσουμε κάτι που υπάρχει ήδη. Έχουμε την Γενική Διευθύνση Ανταγωνιστικότητας που έχει εγκρίνει κάποιες αποφάσεις. Έχουμε πολυμερείς αποφάσεις σχετικά με τιμές, αλλά αυτό αποτελεί δημιουργία καρτέλ. Δεν μιλούμε για ελεύθερη πρόσβαση, αλλά για δίκαιη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Και όλα τα στοιχεία μας δείχνουν, δείχνω εδώ στο slide ένα σημείο, συχνά οι εναλλακτικοί παροχοί δεν έχουν πρόσβαση και προσπαθούμε να το διορθώσουμε αυτό βάζοντας στον κανονισμό αυτό που θα έπρεπε να γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτό δεν είναι παρά η διαφάνεια της σύνοψης που δείχνει την επεμβατική λογική, το πράσινο τμήμα, πράσινο είναι το χρώμα της ελπίδας, θέλουμε αποδοτικές, αποτελεσματικές αγορές, να αντιμετωπίσουμε ζητήματα της δύναμης της αγοράς, ασυμμετρίες, στο δεύτερο πλαίσιο έχουμε τις πρόσθετες τιμές για ευάλωτους πελάτες. Το μεγάλο κόκκινο πλαίσιο δείχνει τους εθνικούς ρυθμιστές, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν ζητούμε πρόσθετες εξουσίες για την Επιτροπή. Εδώ ισχύει η επικουρικότητα, οι τοπικές αγορές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, όπως και οι λύσεις. Αλλά χρειάζονται όλοι τους περισσότερες πληροφορίες για να κάνουν αυτό που αναφέρεται στο μπλε πλαίσιο, να παρακολουθήσουν, να επιτηρήσουν τις αγορές όταν ο ανταγωνισμός δεν αποδίδει αυτό που θα έπρεπε, όταν το υφιστάμενο δίκαιο δεν επαρκεί, όσον αφορά την αποστολή δεμάτων, για να δούμε κατά πόσον οι προϋποθέσεις για την αποστολή δεμάτων εφαρμόζονται κατάλληλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Um, Πρόεδρος, έχω κάποιες ερωτήσεις. Κάλλας, Χωσέ, Άντερσον, Ντίτα, Τζούλια, Ρόζα, Άλγα και εγώ. Σύντομες ερωτήσεις, παρακαλώ. παρακαλώ. Καλώς. Ευχαριστώ. Έχω πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το γεωγραφικό αποκλεισμό. Ο κανονισμός αυτός απαγορεύει τις διακρίσεις εξαιτία ε, μεθόδων πληρωμών. Σε πολλές συναλλαγές όμως η δικαιολογία είναι ο αριθμός του τηλεφώνου. Δηλαδή, στις περιπτώσεις μεταφοράς χρειάζεται ένα τηλέφωνο για να ειδοποιηθεί ο πελάτης και δεν δέχεται το σύστημα ξένα νούμερα ούτε καν για διευκόλυνση στο help test. Αυτή η διάκριση που βασίζεται στον αριθμό του τηλεφώνου πώς αντιμετωπίζεται από τον κανονισμό. Επίσης για τις μεταφορές. κατάλαβα ότι η εξαίρεση για τις υπηρεσίες όσον αφορά τις μεταφορές υπάρχει επειδή υπάρχει το REFIT. Τα δικαιώματα των επιβατών σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους επιβάτες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχει γεωγραφικός υποκλεισμός και δεν μπορεί να κάνει την παραγγελία του όπου θέλει ο πελάτης. Και όσον αφορά την άρνηση επίδοσης, νομίζω ότι και αυτή την πρακτική του γεωγραφικού αποκλεισμού θα πρέπει να τη δούμε πιο πολύ. Έχει να κάνει με την αποστολή των δεμάτων επίσης δηλαδή ο γεωγραφικός αποκλεισμός και η αποστολή των δεμάτων είναι συνδεδεμένα. Όταν διαβάζω την ε, πρόταση, σκέφτομαι τις περιπτώσεις Για παράδειγμα, όλες αυτές οι startups και όλες αυτές οι νέες ιδέες για την αποστολή δεμάτων. Πολλές φορές το άχθος είναι πολύ μεγάλο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να καταγραφούν. Είπατε επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι στη χώρα μέλος. Δηλαδή αν καταγραφεί σε μια χώρα μέλος αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αποστείλει σε όλες. Όχι όμως γιατί η πρόταση λέει ότι οι χώρες μέλη θα συγκεντρώσουν τις πληροφορίες. Δηλαδή σε όλες τις χώρες μέλη πρέπει να καταγραφεί η επιχείρησή σου για να μπορείς και να αποστέλεις δέματα εκεί. Για τις επιχειρήσεις που δίνουν πληροφορίες, μία φορά από ό,τι έχω καταλάβει. Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε άλλες γενικές διευθύνσεις όσον αφορά την ενιαία ηλεκτρονική ψηφιακή πύλη οι τιμές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής υπάρχει κάποια σχέση. Θα είναι open data, ανοιχτά δεδομένα, θα μπορούν δηλαδή να ξαναχρησιμοποιηθούν για τις επιχειρήσεις. Μήπως δημιουργούμε επιπλέον βάρος με την ομοθεσία αυτή. Αξιολογώντας τώρα το κόστος, τις τιμές, μου θυμίζει σαν να πρόκειται για ρύθμιση τιμών εδώ. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το καθορισμό της τιμής, γι' αυτό τι κάνουμε. Οι επιχειρήσεις ίσως θα μπορούσαν να δίνουν περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές για τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουν στην τιμολόγησή τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να επικεντρωθεί όχι στο θέμα της διάρθρωσης της τιμολόγησης, αλλά σε, στο κόστος μόνο. Θέλω και εγώ να ρωτήσω κάποια πράγματα για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, λέει κυρία Ροζιέρ. Στα παραδείγματα που μας δώσατε, όλα βρίσκουν λύση χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ρύθμιση με την, υπηρεσία, με την οδηγία για τις υπηρεσίες δηλαδή φτάνει. Γιατί τώρα να έχουμε κάτι παραπάνω. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι με έπεισε η απάντηση που δώσατε σε αυτό μέχρι τώρα. Έπειτα το πεδίο εφαρμογή. Ακούσαμε ότι για τα οπτικοακουστικά για παράδειγμα εξαιρούνται, είναι εκτός. Ενώ για τα καταλήματα αυτά καλύπτονται εδώ. Τι γίνεται λοιπόν με κάποιον ο οποίος ε, θεωρείται το YouTube το οποίο κανονικά έχει και τα δύο. Τι εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση, θα εφαρμόζω όταν ο κανονισμός. Αναρωτιέμαι επίσης για τα κριτήρια του άρθρου 2, εκείνα που λένε ότι μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση αν η χώρα του πολιτή, του παρόχου και του καταναλωτή, αν η χώρα είναι ίδια, αλλά είναι διαφορετική υπηκότητας. Μα και τότε δεν έχουμε διάκριση βάσει της υπηκότητας σε αυτή την περίπτωση, κάτι το οποίο αντιβαίνει σε όλες τις αρχές της λειτουργίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τη σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες, αν έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες και η τοποθεσία παροχής των υπηρεσιών δεν καθορίζεται γιατί είναι εξ αποστάσεως. Πραγματογνωμοσύνη, νομική, οικονομική για παράδειγμα. ο κανονισμός υπερέχει της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Οπότε τι γίνεται με την αρχή προέλευσης. Και αυτή τη μεγάλη συζήτηση που είχαμε και για τις οδηγίες, την οδηγία για τις υπηρεσίες. Και τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η διάρθρωση ανάμεσα στο γεωγραφικό αποκλεισμό και τον κανονισμό Ρώμη 1. Η Ρώμη 1 είναι κάτω από τον κανονισμό και αυτό τι σημαίνει τότε για την προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Άντερσον, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτό το οποίο γίνεται τώρα και πρέπει να γίνει. Κάποιες ερωτήσεις έχω. Πρώτον για τις λεπτομέρειες για τα άρθρα όσον αφορά τα στοιχεία που θα συλλέγονται πληροφοριακά. Δεδομένης της ομολογίας για το έργο της Επιτροπής που έγινε για την κατάσταση όσον αφορά θέματα απασχόλησης, ε, περιπτώσεις. Ε, Δεν θα έπρεπε η, το θέμα των δεμάτων διασυνοριακά και η παράδοσή τους ε, να συνοδεύεται με περισσότερα στοιχεία γιατί για τους παρόχους και τον αριθμό ατόμων που εργάζονται. Θέλουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να αξιολογούμε την αγορά παράδοσης δεμάτων. Πρέπει να ξέρουμε σε σχέση με τις ώρες απασχόλησης ε, για την παράδοση και συναφή θέματα τι συμβαίνει. Και σε ένα συναφές θέμα, όταν υπάρχει μια τέτοια πρόταση, ο τρόπος υποβολής αυτών των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Εδώ και πολλά χρόνια τώρα έχοντας αυτή την κατάσταση δεν είμαι σίγουρη ότι θα θέλαμε μια τέτοια λύση. Ενώ ακούγεται τεχνικού χαρακτήρα αυτού του είδους τα στοιχεία θα ήταν κάτι που θα θέλαμε πολύ πιο προσεκτικά να εξεταστούν και με τον τρόπο συλλογής τους ε, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας επ' αυτού και για τους στόχους ε, για την ε, διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών όλων δηλαδή των στόχων των καθολικών υπηρεσιών πανευρωπαϊκά δεν θα έπρεπε να έχουμε ιδιαίτερα για την προσπελασιμότητα την προς, προσβασιμότητα, κάποια κάποιας εξειδικευμένα στοιχεία και μια γενικότερη αναστοχαστική παρατήρηση. Κατανοώ βέβαια την ανάγκη της επικουρικότητας, αλλά σχεδόν φαίνεται ότι θα θέλετε να κάνετε περισσότερα, αλλά λέτε ότι πρέπει να επαφεθεί το θέμα στις ρυθμιστικές εθνικές αρχές. Κάποιες από αυτές είναι πολύ καλύτερες από άλλες σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Δεν αληθεύει ότι αν είχατε την ελευθερία δράσης ε, εσεί ε, θα μπορούσατε να κάνατε περισσότερα εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τομέα αντί να δώσετε όλα τα δικαιοδοτικά αυτά ε, δικαιώματα σε ρυθμιστικές αρχέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση που έκανε. Και πράγματι είχαμε μια πρώτη συζήτηση σε αυτό το πακέτο και για τα ψηφιακά με την κυρία Τζούροβα σήμερα το πρωί και κάποιες αψερωτήσεις έχουν απαντηθεί, αλλά κάποια απάντηση απουσιάζει σε σχέση με την ε, επιμεριστική οικονομία, για παράδειγμα. Μας αρέσει η πρότασή σας, ταυτόχρονα όμως διαβάζουμε σε δημοσιεύματα τι γίνεται σε σχέση με κάποια κράτη-μέλη. Θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε με αυτό το χατοφυλάκιο το δυνατόν γοργότερα και να υιοθετηθεί, να διασφαλιστεί η ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι κατακαιρματισμένα 28 διαφορετικές πρωτοβουλίες ή προσεγγίσεις. Λοιπόν, η παρέμβασή μου, η ερώτησή μου. Θα ήθελα να ξέρω πότε ακριβώς θα προβλεφθούν και θα διατεθούν οι κατευθυντήριε γραμμές προς αυτές, για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή και εγώ, λέει η κυρία Ρέντα, για την εισαγωγή παρουσίαση των νέων προτάσεων. Μια ερώτηση για τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Αν κατανόησα την Επιτροπή σωστά, δικαιολογήσατε την ανάγκη ε, μιας νομοθετικής ρύθμισης επειδή οι οδηγίες για την επιβολή του άρθρου 22 της οδηγίας περιπηρεσιών δεν πέτυχε τα ευκαιρία αποτελέσματα. Τα κράτη-μέλη δεν άλλαξαν, δεν τροποποίησαν τις ε, νομοθεσίες τους, τα νομοθετικά τους πλαίσια αντίστοιχα. Για το θέμα των κατευθυντηριών γραμμών είπατε για το ψηφιακό περιεχόμενο. Το μόνο αντικειμενικό κριτήριο είναι αν θα έχει ή όχι ε, μια άδεια για αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο ο πάροχος. Γιατί λοιπόν για το γεωγραφικό αποκλεισμό <clears throat> δεν ε, έχουμε και το θέμα του ψηφιακού περιεχομένου ακόμα και όταν ε, έχει μια τέτοια άδεια ο πάροχος. Από ό,τι γνωρίζω δεν θα υπάρχει τρόπος μέσα στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης copyright πνευματικών δικαιωμάτων να ενταφεί αυτό, διότι δεν είναι θέμα ε, δικαιωμάτων ή copyright. Δεν θα έπρεπε η ρύθμιση αυτή να αντιμετωπίζει το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού σε σχέση με το άρθρο 22 και τις υπηρεσίες ε, Διαρωτώ με ποια, θα είναι, ποια είναι η διαφορά. Αν προσφέρουν οι παιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια ή μουσικά, μουσική ως περιεχόμενο, αν ε, σε σχέση με τα ε, ζητήματα τα οποία αφορούν την ε, νομοθεσία copyright γιατί γίνεται αυτό. Είναι επειδή ε, υπάρχουν κάποια αντικειμενικοί λόγοι για να γίνεται μια τέτοια διαφοροποίηση. Γνωρίζω ότι αναφέρατε επίσης στην πρόταση ότι στην αναθεώρηση, στην επανεξέταση θα εξετάσετε αν θα συμπεριλάβετε το ψηφιακό περιεχόμενο στο μέλλον. Θα ήθελα να γνωρίσω πρώτα απ' όλα γιατί γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Αν το copyright δεν είναι ο λόγος για αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι σαφές ότι σε σχέση με τους καταναλωτές ε, δεν υπάρχει η ανησυχία αυτή. Ωστόσο το ψηφιακό περιεχόμενο είναι στον πυρήνα, στην καρδιά του προβλήματος ε, και ίσως σε σχέση με το γεωγραφικό αποκλεισμό ε, μπορεί κανεί να διαπιστώσει ότι οι άδειε είναι πράγματι ο λόγο. Θα ήθελα να κατανοήσω Ποιο είναι ο λόγο και γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στην νομοθετική αυτή ρύθμιση. Ευχαριστώ. Eh, eh, Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση πρώτα για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Χαιρετίζω αυτή την πρόταση πρέπει να πω σήμερα με την κυρία Επίτροπο Γιούροβα συζητήσαμε και επιθυμούμε να υπάρχει μια επέκταση ώστε να καλύπτεται και το θέμα των γεωγραφικών αποκλεισμών. Είχαμε επίσης και την προσέγγιση ή την έννοια της ευρύτερης, ε, των ευρύτερων παραβάσεων και παραβιάσεων Πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές και έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρξουν αυστηρά κριτήρια τα οποία θα ισχύουν και θα είναι σεβαστά. Τώρα, σε σχέση με τη συνεργασία των ε, εποπτικών αρχών και ρυθμιστικών αρχών θα ήταν πολύ σημαντική υπόθεση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα εδώ και υπάρχουν και περιφερειακές ιδιομορφίες ε, και ιδιαιτερότητες που καθιστούν αυτή τη συνεργασία ευκταία. Ευχαριστώ. Um, thank Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Φυσικά πολύ προσεκτικά, ναι, η κυρία Τούν Χόινστάιν, θα αναλύσουμε τα θέματα αυτά των καταναλωτών. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε. Τώρα υπάρχουν στις προτάσεις σας αυτές και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων για αυτές τις προτάσεις. Θα ήθελα εδώ σε ένα θέμα να επιμείνω. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια υποχρέωση για πωλήσει. Δεν υπάρχει υποχρέωση για πωλήσει. Υπάρχει όμως υποχρέωση να υφίστανται ενιαίες τιμές, οι ίδιες τιμές δεδομένων κάποιων καταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διερωτώ με η άρνηση πώληση. Ε, είναι χειρότερη κατάσταση δημιουργεί για τον καταναλωτή από ότι οι διαφορετικές τιμές ή οι πιο ακριβές τιμές δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με διαφοροποιημένο τρόπο αντιστρέφοντας τους όρους αυτή την κατάσταση. Και πρέπει να πω ότι πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα πολλές πτυχές αυτής της πρότασης ε, για την παράδοση δεμάτων και με το, το γεωγραφικό αποκλεισμό συνδέεται στενά το θέμα της παράδοσης δεμάτων διασυνοριακά. Πρέπει να το δούμε λοιπόν, να έχουν πρόσβαση σε υποδομές και να υπάρχει καλύτερη εποπτεία για τους ε, μικρούς επιχειρηματίες που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει έτσι πραγματικά να εργαστούμε ώστε να υπάρξουν οι αναγκές αλλαγές ε, προς όφελός τους. Και δύο λόγια ίσως ε, προς την κυρία Ρέντα, νομίζω θα συμφωνούσατε μαζί μου ότι θα έπρεπε να αναλυθούν ίσως οι όροι, θα έπρεπε να συζητήσουμε την διεύρυνση, την επέκταση αυτού του φάσματος των θεμάτων ψηφιακού περιεχομένου για το οποίο κάνατε λόγο και θα έπρεπε να αναλώσουμε και κάποιο χρόνο προβληματιζόμενοι από αυτόν. Ευχαριστώ. Um, I've δύο ερωτήσεις. Μία για το γεωγραφικό αποκλεισμό και μία για την αποστολή δεμάτων και είμαι σίγουρη πως θα έχω πολύ περισσότερες, αλλά για τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Είπαμε κάτι πολύ ξεκάθαρο, πως ένας ειδικευμένος έμπορος δεν θα πρέπει να ξαναγκάζεται να πωλεί σε πελάτες εκτός του, της τοπικής του περιοχής, αν δεν το θέλει. Στην πρόταση για το γεωγραφικό αποκλεισμό λέτε πως δεν πρέπει να παραδώσετε να στείλετε σε έναν πελάτη σε μια άλλη χώρα, αλλά θα πρέπει να τους... θα πρέπει να δεχτείτε παραγγελίες. Αυτό που γίνεται με τους πολιτές εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, το ζήτημα είναι ποιος νόμος περί ότι ισχύει, εφαρμόζεται και σε ποια περίπτωση θα βρεθούν σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να δραστηριοποιούνται με 20 διαφορετικές εθ, εθνικές νομοθεσίες. Αυτό προκαλεί σύγχυση στους λιανοπολιτές. Γι' αυτό και υπάρχει η ανησυχία πως οι μικροί λιανοπολιτές απλά μόνο δεν θα, δεν θα προσφέρουν προϊόντα στο διαδικτύο. Αυτό που βλέπουμε είναι πως δημιουργείται σύγχυση, δυσκολίες και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι για αυτόν τον λόγο αποσύρουν τα προϊόντα τους από την προσφορά. Γι' αυτό και πιστεύω πως εάν δεν το κάνουμε σωστά, πιστεύω ότι θα χάσουμε τους μικρούς λιανοπολιτές. Και από ό,τι φαίνεται εντός της πρότασης υπάρχει σύγχυση σχετικά με το πιο δίκαιο περί καταναλωτών ισχύει. Όταν πουλάει κανείς εξ αποστάσεως. Το δεύτερο ζήτημα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Έχει να κάνει με το ζήτημα της ταχυδρομικής αποστολής δεμάτων. Από ό,τι κατάλαβα, εάν εισάγεται αγαθά τις ομένες χώρες και το κάνετε μέσω δέματος και όχι πακέτου, δηλαδή ένα, που είναι ένα μικρότερο, λίγο μικρότερο αντικείμενο, τότε μπορείτε παραδείγματο χάρη να εισάγετε από μια αναπτυσσόμενη χώρα, παραδείγματο χάρη από την Κίνα, μεγάλο αριθμό αγαθών, να τα αποθηκεύσετε παραδείγματο χάρη στη Γερμανία και στη συνέχεια να τα διανύμετε σε όλη την Ευρώπη με πολύ χαμηλότερα έξοδα αποστολή. Εάν ήσασταν ένας Ευρωπαίος πολιτή. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε ανταγωνισμό μέσα στι προποθέσει. Γι' αυτό βλέπω πως τα έξοδα αποστολή είναι πολύ ψηλότερα σε κάποιες χώρες επειδή χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση της αδικίας αυτής ότι υπάρχει δυνατότητα φτηνότερης αποστολή δεμάτων ή πακέτων. Ασχοληθήκατε με το ζήτημα αυτό. Είναι ζήτημα άδικου ανταγωνισμού επειδή κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξαίρεση αυτή των πακέτων ενώ άλλοι όχι. Ευχαριστώ πολύ. those are all... Πιστεύω αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές για τις σημαντικές ερωτήσεις που θέσατε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ομάδες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω πως τα κίνητρα, η πρόθεση της Κομισιόν πίσω από τη δέσμη μέτρων είναι να δώσει στους καταναλωτές περισσότερες δυνατότητες επιλογής και περισσότερες ενδιαφέρουσες προσφορές. Αλλά βασική πρόθεση της Επιτροπής είναι επίσης πως δεν θα προσθέσουμε και άλλα εμπόδια για τους εμπόρους. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη νομική βεβαιότητα μπορούμε για τους εμπόρους. Και αυτό είναι σημαντικό. Επειδή διάφορα, διάφορα μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για φραγμούς που ίσως δημιουργηθούν από το μέτρο αυτό. Yes, Επίσης θα ήθελα να πω πως ελπίζουμε να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο στο ζήτημα της παράδοσης ζεμάτων, αλλά εδώ τώρα αναφερόμαστε σε καταστάσεις που δεν επηρεάζονται από την αποστολή δεμάτων. Ακόμη και χωρί την αποστολή δεμάτων, θα υπάρχουν οι έμποροι που θα ήθελαν να κατακαιρματίσουν η αγορά. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να πούμε πως να περιμένουμε μέχρι να εφαρμοστούν όλα τα άλλα μέτρα. Επειδή δεν σχετίζονται με αντικειμενικούς λόγους διακρίσεων, όπως έχουμε στην αποστολή δεμάτων ή στον περίπλοκο χαρακτήρα του εφαρμοστέου δικαίου. Και πάλι όπως είπα, 8 25% των συναλλαγών πλήττονται από αυτόν. Λοιπόν, για το εύρος τώρα, αποκλείουμε κάποιες υπηρεσίες. Στον τομέα των μεταφορών, οι μη διακρίσεις ήδη έχουν ενσωματωθεί σε ένα μεγάλο αριθμό σχετικονομικών κειμένων, ιδίως στα αεροπορικά ταξίδια και στα επίγεια και θαλάσσια ταξίδια, αλλά όχι ακόμα στα σιδηροδρομικά εκεί η αρχή που δεν πρέπει να χρεώνεται διαφορετική τιμή επειδή παραγγέλνει κανείς ένα εισιτήριο από ένα άλλο κράτο μέλος ήδη εφαρμόζεται με την εξαίρεση των σιδηροδρομικών ταξιδιών όπου η Κομισιόν θα κάνει μια πρόταση του επόμενου μήνε. Όσον αφορά τα οπτικοακουστικά και το υλικό που προστατεύεται από copyright θα ασχοληθούμε με τον, στα πλαίσια του εξυγχρονισμού του copyright με την προώθηση της μεγαλύτερης πρόσβασης σε ακουστικά αντικείμενα περιεχόμενα. Καλύπτουμε περιεχόμενα μη οπτικο-ακουστικού χαρακτήρα που προστατεύονται από copyright. Δεν εφαρμόζουμε, εκτελούμε το άρθρο 4 σχετικά με αυτό, είναι το άρθρο που ορίζει την έλλειψη διακρίσεων. Ο λόγος γι' αυτό είναι πως την αξιολόγηση αντικτύπου δεν είχαμε επαρκείς πληροφορίες για να αξιολογήσουμε εάν θα υπάρξουν ανθέμητες συνέπειες. Τώρα μιλούμε για μουσική και ηλεκτρονικά βιβλία, είναι ιδιαίτερες αγορές και στον τομέα της μουσικής ο κανόνας είναι πως υπάρχουν ευρωπαϊκές άδειες. Αλλά αυτό δεν ισχύει κατά 100% επειδή υπάρχουν καταστάσεις όπου ακόμη και μεγάλοι παροχής όπως το Spotify προσφέρουν μουσική για την οποία εμείς θεωρούμε πως δεν κατέχουν άδεια. Γι' αυτό πολλές φορές ένας χρήστης μπορεί να ζητά μια υπηρεσία και αυτή η υπηρεσία να μην διατίθεται στον καταναλωτή επειδή αυτή δεν καλύπτεται από το Εθνικό Δίκαιο Αδειοδότησης. Στον τομέα των ηλεκτρονικών βιβλίων κάποια κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία που ορίζει σταθερές τιμές και η οποία είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό και αν πωλείται ηλεκτρονικά βιβλία σε ένα κράτο μέλος το οποίο έχει με τέτοια νομοθεσία σταθερών τιμών θα πρέπει να χρεώσετε για το βιβλίο στη γλώσσα της χώρας αυτής την τιμή που ορίζεται ως σταθερή τιμή βιβλίου στη χώρα αυτή. Αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, ιδίως αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση, επειδή πρέπει να βρείτε ποια είναι η κατάλληλη τιμή, η τιμή για οποιαδήποτε βιβλίο στην κάμα σας. Γι' αυτό και εδώ δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ποιο θα ήταν ο διοικητικός φρα... φραγμός, ο γραφειοκρατικός φραγμός για τους πολιτές βιβλίων. Όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο, η Συμφωνία Ρωμή 1 βρίσκεται σε ισχύ. Τώρα, είτε εφαρμόζεται ή όχι το δίκαιο περί καταναλωτών, εξαρτάται από την κατάσταση στην εκάστοτε ε, συγγνώμη. Τι, τι ακριβώς είπατε, είπα... Διευθύνω. Έχετε τη δυνατότητα να διευθύνετε τις δραστηριότητές σας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Και γι' αυτό θα έχετε πληροφορίες στην ιστοσελίδα σας, στη γλώσσα του καταναλωτή, θα έχετε διευθύνσεις. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα καθορίσουν κατά πόσον η εταιρεία απευθύνεται ή όχι στη χώρα αυτή. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με την απόκριση μιας εταιρείας, ιδίως όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός περί γεωγραφικού αποκλεισμού, ιδίως όσον αφορά την πώληση υπηρεσιών και αγαθών. Είναι πολύ πιθανόν ο καταναλωτής να, να μην ζει στη χώρα στην οποία απευθύνεται, διευθύνει ο πολιτής. Και σε αυτή την περίπτωση όμως η Συμφωνία Ρώμη 1 δεν επηρεάζεται επειδή ο πολιτής δεν απευθύνεται στο, στη συγκεκριμένη χώρα. Και γι' αυτό ο καταναλωτής προσεγγίζοντας την ιστοσελίδα αυτή με την ελευθερία που δίνει ο κανονισμός περί γεωγραφικού αποκλεισμού, ζητά για την παροχή μιας υπηρεσίας η οποία διέπεται από το δίκαιο του εμπόρου. Αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από την κατάσταση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ρώμη 1. Εκεί πρέπει να οριστεί, ο πολιτής πρέπει να ορίσει ακριβώς την γεωγραφική, γεωγραφική περιοχή στην οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί εμπορικά. Εκεί ο πολιτής απευθύνεται σαφώς και αποκλειστικά στο κράτος μέλος Α ή Β και αν ο πολίτης και αν ο πελάτης προέρχεται από ένα άλλο κράτος μέλος, τότε ο πολιτής θα καθορίσει κατά πόσο ισχύουν οι κανόνες. Επίση υπάρχει παραδείγματο χάρη το ζήτημα κατά πόσον μέσω ενός τηλεφώνου ο πολιτή θα απαντήσει και σε ποια γλώσσα στον πελάτη. Όμω ο πολιτή δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει υπηρεσίες στη γλώσσα του πελάτη. Εδώ η προσέγγιση είναι αυτή τη μεταχείρισης. Δεν θα μεταχειριστείτε χειρότερα, αλλά ούτε και καλύτερα θα λάβετε μεταχείριση αν παραγγείλετε από μια σελίδα στη Γερμανία θα επικοινωνήσετε στα γερμανικά. Είναι παρόμοιο με τον πραγματικό κόσμο. Αν πάτε στη Γερμανία και αγοράσετε κάτι από ένα κατάστημα θα μιλήσετε στα γερμανικά. Δεν υπάρχει καμία αποχρέωση πώληση. Είναι μια μικρή διαφορά. Αλλά υπάρχει μια αποχρέωση μη διακρίσεων οι περισσότερε εταιρείε έχουν την ελευθερία να μην πολλούν για πολλού λόγου. σω έχουν μείνει από αποθέματα ή έχουν προϊόντα που απευθύνονται σε πελάτε πάνω από ένα όριο ηλικία. Αλλά αν έχετε μια άλλη εθνικότητα, προέρχεστε από ένα άλλο κράτο μέλος, κράτος μέλος, τότε υπάρχει μια υποχρέωση να μην προβαίνουν επιχειρήσεις σε διακρίσεις. Εδώ έχουμε εντοπίσει πέντε καταστάσεις συγκεκριμένες για τις οποίες η νομοθεσία αναφέρει πως είναι περιπτώσεις αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού. Το νομοθετικό πλαίσιο συνεχίζει να ισχύει, αλλά στο πλαίσιο των συναλλαγών αυτών υπάρχουν πέντε συναλλαγές στις οποίες δεν είναι πλέον δικαιολογημένος ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Πρόκειται δηλαδή για μια συμπλήρωση της οδηγίας περί υπηρεσιών. Αυτό δεν αφορά την κατάσταση στη χώρα προέλευσης από την οπτική γωνία του εμπόρου. Εδώ αναφερόμαστε στην οπτική γωνία του πελάτη που προσπαθεί να ασκήσει το δικαίωμά του σε, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ένα λεπτό καθένας. Για να είμαστε εντελώς ξεκάθαροι, ο κανονισμός αυτός δεν έχει να κάνει τίποτα με τη χώρα προέλευσης. Εδώ πέρα μιλάμε για τους κατανολητές που πάνε αλλού, ενώ χώρα προέλευσης έχει να κάνει με τον έμπορο ο οποίος αλλάζει χώρα. Δεν είμαστε σε αυτή τη λογική όμως, για να είναι ξεκάθαρο το θέμα. Πρόεδρος παρακαλώ. Θέλω και εγώ να εξηγήσω ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στον άρθρο 16, όπου υπάρχει πολλή ελαστικότητα. Είναι μια συντονισμένη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χώρες μπορούν να μας ζητήσουν το συντονισμό. Υπάρχει δυνατότητα βάση του κανονισμού, αλλά τώρα ξεκαθαρίζεται ακόμα περισσότερο και υπάρχει και νομική βάση. Η νέα δυνατότητα να αναλάβει την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια δράση απαιτεί τα τρία τέταρτα ε, του πληθυσμού και των χωρών μελών. Αυτό το έχουμε δανειστεί από άλλες αντίστοιχες πολιτικές συμμόρφωσης γιατί θέλαμε να έχουμε σαφή κριτήρια για το πότε μπορεί να αναλάβει αυτό τον ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σημαίνει ευρεία παράβαση. Πότε μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το συντονισμό η ευελιξία είναι μεγαλύτερη. Έχουμε τις περιφερειακές αρχές ναι, και μπορούμε να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές ε, συμμόρφωσης, ώστε αυτές να μπορούν να συνονούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, εσείς. Όσον αφορά το διοικητικό άκθος, σίγουρα για τις startups, ε, ναι, αλλά υπάρχει ένα όριο για να αποκλείονται κάποιες ε, μικρές επιχειρήσεις, γιατί εδώ πέρα θέλουμε να διευκολύνουμε την κατάσταση και με την επιτροπολογία. Οι ρυθμιστές πολλές φορές ζητούν πληροφορίες με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ε, νομίζω εδώ πέρα θέλαμε μία μόνο μορφή που να ικανοποιεί και τις 28 χώρες. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει ε, βελτίωση για τις τιμές. Μιλάμε για 15 τιμές που επιλέγουμε που έχουν να κάνουν με το εμπερικό, με το ηλεκτρονικό εμπόριο. δεν χρησιμοποιούνται κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας και αυτό έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο naming and shaming. Υπογραμμίζουμε ότι πρέπει οι ρυθμιστές να κάνουν τη δουλειά του. Συμπληρώνουμε την ταχυδρομική οδηγία. λέμε ότι πρέπει να είναι προσιτό το κόστος. Θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει μια διαφορετική ονομασία. Μας ενδιαφέρει η δομή της τιμής. Να καταλάβουμε γιατί τους αναγκάζουμε να μας πούνε. Και αν δεν μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί πολλαπλασιάζουν επί 10 την τιμή εκτός της χώρας όπου βρίσκονται, ε, θα αναγκαστούν να το ξανασκεφτούν και ίσως να μην το κάνουν. Τώρα ναι, ό,τι πληροφορίες θέλατε θα μπορούσατε να προσθέσετε στον κατάλογο, αλλά τότε αυτό θα ερχόταν σε αντίφαση με αυτά που είπαμε πριν για την απλοποίηση. Γι' αυτό περιλαμβάνουμε μόνο ό,τι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε την αγορά. Δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Το άρθρο αυτό όμως επιδέχεται συζήτηση προσβασιμότητα τώρα, πέρα από το προσιτό της τιμής. Και εδώ στην οδηγία για τα ταχυδρομεία υπάρχουν ε, πολλά για περιθώριο στον εθνικό ρυθμιστή νομοθέτη να το κοιτάξει. Τώρα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Εδώ μιλάμε για μία, ε, ένα έντυπο που θα συμπληρώνει το άρθρο 3 όλες οι παράμετροι πρέπει να αναφέρονται στο άρθρο 3 και εκεί είναι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει τη σοφία του και τα δικαιώματά του. Η εφαρμοστική πράξη θεωρούμε ότι είναι το καταλληλότερο μέσο. Για το UPU πακέτο. Φυσικά, το γνωρίζουμε, ναι, υπάρχει. Και αυτό ακριβώ είναι που δείχνει τη δυσκολία. Είναι υποχρέωση που απορρέουν από τη διεθνή νομοθεσία. Υπήρξε ένα ε, συνέδριο πρόσφατα και του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη. Από το 92 προσπαθούν να βρουν λύσεις οι χώρες. Πολλές προτάσεις υπάρχουν για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και διμερώς ανάμεσα στα ταχυδρομεία υπάρχουν ε, συνεννοήσεις στο UPU. Ναι, προσφέρει υπηρεσίες και στους Κινέζους. Και οι Κινέζοι ενδιαφέρονται, αλλά θέλουν να υπάρχουν ίχνη. Οπότε μπορεί να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην έλλειψη ισοτιμίας με τις εισαγωγικά αναπτυσσόμενες χώρες. Οι υψηλές τιμές αντισταθμίζουν ακριβώς αυτό. Απ' τη μια οι τιμές παραδοσιακά ήταν υψηλές και πολύ πριν τους παίκτες Κίνα και λοιπά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές, 32 λίρες για ένα κιλό για παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς δεν πουλάνε πολύ κανένας, δεν θα πληρώσει για ένα τέτοιο πακέτο. Ακριβώς γι' αυτό και οι πιο ολιανικοί δεν θα πουλήσουν τέτοια προϊόντα. Θέλουμε μια αποστολή να μπορούν να αναπτύξουν το εμπόριό τους. Θέλουμε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη φύρμα τους επιχειρήσεις αυτές ακριβώς για να βελτιώνεται οι δραστηριότητές τους και να γίνονται πιο γνωστοί στην αγορά. Ευχαριστούμε. Τώρα έχουμε τους νέους κανόνες για τα οπτικοακουστικά. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης θα δώσω το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποιον? Λορένα Βοσακλόντσο. Εσείς, Λορίνα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Διότι βρίσκεστε εδώ επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήδη. Λοιπόν, για την παρουσίαση, επεξήγηση. Ναι, με βλέπετε εδώ. Την φιλοσοφία που εμπνέει, που διέπει αυτή την πρόταση. Να ανέβω εκεί, να έρθω σε εσά, εντάξει. So, uh, the philosophy... Εντάξει λοιπόν, για την φιλοσοφία που μας ενέπνευσε είναι κατά κάποιο τρόπο όπως περιέγραψε ο Επίτροπος Έτινγκερ και από πλευρά δεν είναι μια επανάσταση, είναι μια εξελικτική διαδικασία. Είναι μια οδηγία που υπάρχει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, ούτω ή άλλω. Και η ιδέα που μα ενέπνευσε ήταν να διατηρήσουμε αυτό που λειτουργεί και είναι αποτελεσματικό και για τα υπόλοιπα τμήματα να εξυγχρονίσουμε και να επικαιροποιήσουμε την οδηγία για να είναι πιο αποτελεσματική και να λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά οπτικοακουστικών ώστε να είναι αποτελεσματική. Και έτσι λοιπόν όχι μόνο θα υπάρξει διατήρηση αλλά και ενδυνάμωση, ενίσχυση σε σχέση με τα θέματα ενιαίας εσωτερικής αγοράς και για την ενιαία εσωτερική αγορά σε σχέση με αυτή την οδηγία επιτυγχάνεται με βάση την αρχή της χώρας του κράτους προέλευσης με βάση την αρχή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ότι όσοι εκπέμπουν σε, κάνουν εκπομπές και πάροχοι υπηρεσιών όσον αφορά ε, το Orange ή ε, άλλες εκπομπές πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και κανονισμούς ε, της χώρας αυτής δεν πρέπει λοιπόν να προσαρμόζονται με κανονισμούς 28 διαφορετικών κρατών μελών, αλλά με τους κανονισμούς του κράτους προέλευσης, που λειτουργεί καλά αυτός ο κανόνας ε, και με διαβούλευση και τα συναφή, ώστε σήμερα 38% των διάβλων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λειτουργούν μέσω άλλων ε, χωρών ή στοχεύουν στις ε, χώρες εκπομπών και το ποσοστό που είναι διαθέσιμο στα κράτη, σε κράτη-μέλη προέρχεται από άλλα κράτη-μέλη. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι έχουμε αυτό το ε, πολυσχηδές οποίο στα οπτικοακουστικά. Τι είναι εκείνο το οποίο προτείνουμε τώρα εμείς να γίνει. Φυσικά να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί η αρχή του κράτους προέλευσης και να διευκολυνθεί η λειτουργία του. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα επιτευχθεί. Αφενός η ιδέα είναι να απλουστευθούν οι κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ταυτοποιήσουν και να ανοιχνεύσουν ποια χώρα ε, εκπέμπει μέσω κάποιου παρόχου. Προτείνουμε να υπάρξει διαφάνεια που θα διασφαλιστεί ώστε να μας γνωστοποιούν τα κράτη-μέλη αυτά τα στοιχεία, να υπάρξει μια βάση δεδομένων ποιοι πάροχοι λειτουργούν υπό τη δική τους δικαιοδοσία, ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά οι πάροχοι ποιοι είναι οι ρυθμιστές που είναι αρμόδιοι για αυτούς ώστε να μπορέσουν σε αυτό το πεδίο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Και φυσικά για την αρχή του κράτους προέλευσης η αρχή είναι να πλουστευτεί το πλαίσιο εξαιρέσεων και μηχανισμών παράκαμψης. Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη κατ' να χορηγούν εξαιρέσει σε σχέση με την αρχή του κράτους προέλευσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αλλά οι κανόνες και οι κανονισμοί αυτοί είναι περίπλοκοι και σύνθετοι και είναι διαφορετικοί για την γραμμική, για τις γραμμικές εκπομπές από, από ότι για άλλες ε, εκπομπές. Και με βάση μια συγκεκριμένη λοιπόν διαδικασία για την εξαίρεση θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αυτό. Και για να προαχθεί η διάσταση της εσωτερικής αγοράς σε αυτήν την οδηγία, η ιδέα που είχαμε είναι να γίνει αυτό όχι μέσω περί της ε, εκ του περισσού νομοθεσίας, αλλά να προσεγγίσουμε διαφορετικά ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ενισχύοντας τον ρόλο των ρυθμιστικών αρχών. Αφενός λοιπόν στοχεύουμε προτείνουμε οι απαιτήσει μας να ενταχθούν στην οδηγία ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ένα ή περισσότερους ανεξάρτητους ε, ρυθμιστικούς φορείς ε, ως σώματα και θα πρέπει λοιπόν ε, να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και κριτήρια για να θεωρηθούν ανεξάρτητοι αυτοί οι φορείς και επίσης η πρόταση να επισημοποιηθεί η υφιστάμενη αυτή ομάδα φορέων ρυθμιστικών αρχών στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ομάδα θα αναγνωρίζεται από αυτή την ε, οδηγία και ο ρόλος της ενδυναμώνεται. Η ιδέα είναι να διευκολυνθούν ανταλλαγές μέσω ρυθμιστικών αρχών για την εφαρμογή με το βέλτιστο τρόπο της οδηγίας. Και γι' αυτό λοιπόν προβλέπεται για διάφορα θέματα που είναι ε, μεγάλης εμβέλειας ότι θα μπορούν να διαβουλεύονται ε, οι ρυθμιστικές αυτές αρχές για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή για την ενδυνάμωση της εσωτερικής ε, αγοράς είναι η ενδυνάμωση της αυτορύθμισης. Αυτή η οδηγία λοιπόν μέσω, σε, σε, μεγάλο βαθμό θα βασίζεται στην αυτορύθμιση. Ακόμα και η φύση των παροχών μέσω αυτής της οδηγίας και με την, ε, τα θέματα διαφημίσεων και της προστασίας ε, των ε, ανηλίκων, με την εμπλοκή ρυθμιστικών αρχών στο εθνικό επίπεδο, αυτό που προτείνουμε να είναι να υπάρξουν συγκεκριμένες διατάξεις ώστε αυτή η αυτορύθμιση να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα, να είναι πιο αποτελεσματική. Αλλά ταυτόχρονα επίσης προτείνουμε αν θεωρηθεί ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είναι χρήσιμο, θα υποστηρίζαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ρυθμίσεις ε, που θα μπορούσαν να προαγάγουν ακριβώς την πρόθεση του στόχου της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σε σχέση με τη συνιστόσα της εσωτερικής αγοράς και για την αρχή του κράτους προέλευσης και την ενίσχυση αυτών των συνιστοσών. Από την άλλη πλευρά, όπω έλεγα, ο στόχο μα είναι να εξυγχρονιστεί, να επικαιροποιηθεί αυτή η οδηγία, μια και ισχύει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και τα πράγματα εξελίσσονται ταχύτερα, με ταχύ ρυθμού και μετατίθενται οι καταναλωτές στον ηλεκτρονικό, ας το πω έτσι, ε, στην ηλεκτρονική μέθοδο ε, και διαδικασία ε, συνεννόησης και επαφών στο ηλεκτρονικό πλαίσιο και έχουμε και νέους ε, που εισέρχονται στην αγορά. Ε, κάποιοι ευρωβουλευτές ε, ρωτούσαν σε σχέση με αυτούς τους νέους εμπλεκόμενους που βρίσκονται ή αναφύονται στην αγορά. Εξυγχρονίζοντας τους κανόνες προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις εξελίξεις που σημειώνονται στην αγορά. Καμιά φορά προτείνουμε απορρίθμιση Άλλες φορές προτείνουμε κάποια πράγματα να αριθμιστούν στο εύλογο πλαίσιο όπως χρειάζεται. Για την απορρίθμιση η πρόταση λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι απαιτήσει ε, και οι όροι όσον αφορά διαφημίσεις ε, όταν συσχετίζονται με ένα συγκεκριμένο όγκο διαφημίσεων που εκπέμπονται. Δηλαδή, maximum κατά το μέγιστο 20% ανά ώρα διαφημίσεων αναλύσαμε το ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον και ότι σήμερα δεν είναι αναγκαίο να επιβληθεί αυτός ο περιορισμός στους ε, όσους ε, κάνουν τέτοιες ε, εκπομπές, διότι ήδη με την αυτορύθμιση ρυθμίζουν αυτό το θέμα. Έχουμε νέους εμπλεκόμενους παίκτες στην αγορά, που το θέμα της διαφήμισης δεν είναι τόσο φλέγον. Αν υπάρχει λοιπόν το θέμα της όχι μόνο μπορεί, αλλά και είναι δυνατόν σε πολλές περιπτώσεις ε, λόγω της ε, μεγάλης προσφοράς να προχωρούν χωρίς ε, διαφημίσεις. Να κάνουμε αυτό το πλαίσιο πιο ελαστικό, πιο ευλίγιστο. Αντί να έχουμε το 20% ανά ώρα διαφημίσεων, να έχουμε 20% ημερήσια από συγκεκριμένη ώρα έναρξης μέχρι συγκεκριμένη ώρα λήξης, ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείριση αυτού του, αυτής της αρχής. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει επιβάρυνση ούτως ή άλλως ε, και πίεση από άλλους ε, εμπλεκόμενους εκτός Ευρώπης ε, και να μην είναι γενικόλογοι και αφηρημένοι οι, οι κανόνες και να είναι δυνατόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του θέματος των διαφημίσεων και σε σχέση με τα έσοδα που μπορούν να επιτευχθούν. Να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη ελαστικότητα, μια και δεν είναι πλέον αναγκαίο να είμαστε τόσο αυστηροί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και επίσης ε, με την πρόθεση εξυγχρονισμού των κανόνων προσπαθούμε να πετύχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των κανόνων και κανονισμών σε σχέση με εκείνους που έχουν εκπομπές τηλεοπτικές και ε, τους άλλους παρόχους. Διότι υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις ε, ε, τηλεοπτικές εκπομπές από ότι για τις άλλες παροχές υπηρεσιών. Αν δούμε το θέμα της προστασίας ανηλίκων, Σήμερα το περιεχόμενο, το τηλεοπτικό, ε, πολλές φορές είναι απαγορευτικό για ανήλικους και αν είναι και βλαπτικό ή ε, επιζήμιο πρέπει να υφίστανται περιορισμοί για αυτό. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί αυτό το ε, επιζήμιο περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο και θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να επιβληθούν περιορισμοί. Όμως ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι οι ανήλικοι ε, ενώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας ε, μεγαλύτερης ε, σε σχέση με τέτοιες εκπομπές, ε, η ιδέα μας είναι η προστασία τους να επιτυγχάνεται με τον ίδιο τρόπο για τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά και για τις άλλες παροχές υπηρεσιών ώστε να αυξηθεί το επίπεδο της προστασίας τους για την προαγωγή ευρωπαϊκών έργων ή παραγωγών για τις τηλεοπτικές εκπομπές οι πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν πάνω από το ίμιση του περιεχομένου των εκπομπών με ευρωπαϊκά έργα. Για τις ε, παροχές υπηρεσιών πρέπει να υπάρχει η διάταξη και αυτό ήταν πρόβλημα και έχει και υπήρξαν πραγματικές, ε, πραγματικά προβλήματα και τριβές επειδή δεν υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο ε, για τα παραδείγματα που ε, έχουμε και τον κατακαιρματισμό του τοπίου που υφίσταται τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί να εξευρεθεί μια καλύτερη ισορροπία διότι οι πάροχοι εκπομπών επενδύουν πολύ περισσότερο σε αυτή τη συνιστόσα η ιδέα λοιπόν είναι να διατηρήσουμε τους κανόνες και κανονισμούς ε, για τις ε, τηλεοπτικές εκπομπές ε, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί, να αναβαθμιστεί το επίπεδο των κανονισμών για τις ετούμενες υπηρεσίες. Με ποιο τρόπο σε σχέση με τους κανόνες αυτούς που θα πρέπει να διαμορφωθούν επειδή η λογική παροχής ετούμενων υπηρεσιών δεν είναι, το, δεν είναι η ίδια υπόθεση όπως η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και με πάνω από το 50% ευρωπαϊκών παραγωγών υπάρχει ένας ε, ε, ε, δεσμευτικός περιορισμός. Αν παρακολουθεί κανείς Orange ε, άλλες εκπομπές. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ε, τηλεοπτικά προϊόντα ευρωπαϊκά δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν καλύτερα οι κανόνες αυτοί και να μην είναι τέτοια επιβάρηση για τους παρόχους και να δίνουν και ευδιάκριτο χαρακτήρα στα ευρωπαϊκά έργα, στις ευρωπαϊκές παραγωγές. Φυσικά αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο παρουσίασης ή διάχυσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προϊόντων. Θα πρέπει οι πάροχοι να μπορούν να εκπέμπουν αυτές τις εκπομπές, αλλά να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό έστω 20% που θεωρείται αναλογικό σε σχέση με τον όγκο των όσων εκπέμπονται στην παροχή αυτών των προϊόντων, στην παρουσίασή τους. Η τελευταία πρόταση που έχουμε και κάνουμε για να επικαιροποιηθούν οι κανόνες αυτοί ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της σημερινής εποχής είναι όπως έλεγα πιο πριν υπάρχουν νέοι που έχουν εισαχθεί και εμπλέκονται στην αγορά, νέες πλατφόρμες. Έχουμε εδώ τώρα θέματα οπτικοακουστικών, οπτικοακουστικών πλατφορμών και θα πρέπει να μπορέσουμε να τις λάβουμε υπόψη στις ρυθμίσεις. Είναι πάροχοι που σε διαφορά, σε διαφοροποίηση με τους παρόχους ε, ε, τηλεοπτικών εκπομπών δεν έχουν κάποιον έλεγχο ε, επί της, του περιεχομένου εκπομπών που εκπέμπουν. Βλέπουμε λοιπόν ενώ υπάρχουν κάποιοι που καταναλώνουν περισσότερο το ένα από το άλλο προϊόν και σε σχέση με τους ανήλικους. Η ιδέα και πάλι είναι να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα της αγοράς και να επεκτείνουμε, να διευρύνουμε τους κανόνες και τους κανονισμούς για αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά μόνο εφόσον και κατά τη διάρκεια του διαστήματος που θα είναι αναγκαίο να γίνει αυτό για την προστασία των ανηλίκων και την αναχέτηση των περιορισμών των ε, κηρυγμάτων μίσους, ε, την αναζωπήρωση μίσους ε, και να υπάρξει και η δυνατότητα σε σχέση με την σωστή λογοδοσία να λειτουργήσουν αυτά, ώστε το θέμα της περιορισμένης ευθύνης θα εξακολουθήσει να ε, λειτουργεί, όμως η οδηγία αυτή θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες αυτές να αναλάβουν, να αναλάβουν τα αναγκαία μέτρα για να προστατέψουν τους ε, ανηλίκους από αυτά τα φαινόμενα. Ε, σεβόμενοι την αρχή της περιορισμένης ε, ευθύνης. Η ιδέα είναι ότι οι πάροχοι έχοντας ήδη την προοπτική ανάληψης μέτρων και με την ταχύτερη προέλαση της ε, τεχνολογίας από πλευράς ε, δυνατοτήτων είναι να μπορέσει η ρύθμιση αυτή να λειτουργήσει και με την συμμετοχή και εμπλοκή της ε, ίδιας της βιομηχανίας οπτικοακουστικών. Αυτό θα σήμαινε και σε υστερότερη φάση έναν εναρμονισμό σε σχέση και με τους ε, ε, ρυθμιστές. Αυτές είναι οι προτάσεις μας σε σχέση με την οδηγία. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Julia Rader. Julia Rader. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για την παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα πιστεύω πως είναι καλό που η Επιτροπή δεν αμφισβητεί την χώρα προέλευσης για την παροχή οπτικόπ ακουστικών υπηρεσιών. Αλλά κάποιες ερωτήσεις. Προτείνεται να διαγραφεί το άρθρο. Είπατε πως πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πράξη προσβασιμότητας που θα έρθει. Έχω κάποιο ζήτημα με αυτό. Έχουμε ήδη μια οδηγία περί προσβασιμότητας και εκεί στο τέλος κατόπιν επιθυμίας του Συμβουλίου αποκλείστηκε, αποκλείστηκαν οι, τα, δημόσια κανάλια, οι δημόσιοι σταθμοί. Το ζήτημα είναι ότι η οδηγία ATS θα προχωρήσει μάλλον γρήγορα. Αυτό που είδαμε στην οδηγία περί προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, βλέπουμε πολύ μακρές προθεσμίες εφαρμογής. ακόμη λοιπόν, και αν κατορθώσουμε να συμπεριλάβουμε όλες τις υπηρεσίες στην πράξη προσβασιμότητας, θα, αυτή θα τεθεί σε ισχύ πολύ αργότερα. Θα έχουμε ένα μεσοδιάστημα δηλαδή στο οποίο δεν θα υπάρχει καμία προσβασιμότητα όσον αφορά την συμπερίληψη πλατφορμών μοιρασμού περιεχομένων βίντεο. Γνωρίζουμε το YouTube, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε αυτό. Πιστεύω πως είναι καλό ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα κουμπί αναφοράς με το οποίο μπορούν να αναφερθούν, να αναφερθεί ρητορική μίσους παραδείγματος χάρη. Αν παραδείγματο χάρη πείτε πω είναι μόνο οι πάροχοι που έχουν την συντακτική ευθύνη του βίντεο, αυτό πιστεύω δεν θα ήταν εύλογα εάν κάποιο απλά πουλά χώρο στο διαδίκτυο, στο οποίο κάποιο άλλο μπορεί να ανεβάσει βίντεο. Πώς θα διαφοροποιούσατε τότε που αρχίζει ο όρος πλατφόρμα μοιρασμού περιεχομένου βίντεο και που απλά παρέχεται χώρο στο διαδικτύο. Όσον αφορά το ζήτημα Είπατε ήδη πως δεν μπορείτε να, να συγκρίνετε ένα γραμμικό περιεχόμενο με ένα βίντεο περιεχόμενο. Πιστεύω πως η διάδοση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας είναι σημαντική, αλλά στην πράξη έχουμε το ερώτημα τι είναι ένα έργο. Είμαι πάροχος υπηρεσιών βίντεο λοιπόν και θέλω να έχω μια ποσόσταση 20%. Αρκεί, αρκεί τότε να έχω την άδεια για το Eastlanders που έχει 5.000 επεισόδια. Επίσης όσον αφορά το ερώτημα αυτό, θα ήταν δυνατόν οι πλατφόρμες μοιρασμού βίντεο για να φτάσουν το 20% δεν θα παίρνουν άδειε για νέα, νέες ευρωπαϊκές ταινίες, απλά ότι απλά θα αφαιρέσουν μη ευρωπαϊκές ταινίες. Ποια είναι η θεωρία σας λοιπόν για το πώς η ποσόστοση αυτή στην πραγματικότητα θα προωθήσει το ευρωπαϊκό περιεχόμενο και θα προωθήσει την πολιτισμική μορφή αντί να τη μειώσει. Όσον αφορά τις διαφημίσεις, πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ήδη μια έντονη ρύθμιση σε αντίθεση με, τη, με το διαδίκτυο. Αλλά η κατάσταση στο διαδίκτυο είναι απέσια. Δεν θα πρέπει να εναρμονίσουμε περισσότερο από ό,τι λιγότερο εκεί, το οποίο κάναμε και σε πολλού άλλου τομεί. Όσον αφορά την προστασία ανηλίκων, επίση πρέπει να σκεφτεί κανεί τι διαφορέ του διαδικτύου με του ε, άλλου τομεί. Ένα τρόπο συμμορφώση με τι απαιτήσει προστασία ανηλίκων είναι με τι ώρε, αλλά ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικέ ζώνε ώρα. Μπορούμε να εξετάσουμε δηλαδή εθελοντικέ πρακτικέ τη ε, βιομηχανία, αλλά έχουμε, λέει η πρόεδρο, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Εβελίν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση των προτάσεών σας. Ένα ερώτημα που είχα. Επειδή είπατε προς πρόσβαση σε online πλατφόρμες, την απαντήσατε στο τέλος. Πρόκειται δηλαδή μόνο για τις οπτικοακουστικές πλατφόρμες και όχι πλατφόρμες γενικότερα. Κατά τη διατύπωση της παρουσίασης θα μπορούσε να το κατανοήσει κανείς και διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την αποσαφήνιση. Πιστεύω πως ήταν πολύ σημαντική, επειδή πιστεύω πως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως ταυτόσημες όλες τις πλατφόρμες. Όσον αφορά τα, τις παροχές οπτικοακουστικών υπηρεσιών, συμφωνώ με το ότι πρέπει να ισχύει η αρχή της χώρας προέλευσης. Ίσως ο ένας ή ο άλλος να εκφράσει την απορία του αν ακούσει να μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με το ζήτημα του δικαίου πνευματικών δικαιωμάτων που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο ζήτημα αυτό και πρέπει να λυθεί υπόψη. Εκεί που έχω βάλει ένα ερωτηματικό είναι ο τομέα στον οποίο μιλάτε ανοιχτά για το ότι θέλετε μία απορρίθμιση και μάλιστα στις διαφημίσεις και στην ταξινόμηση των διαφημίσεων των προϊόντων. Ήμουν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη συζήτηση του νόμου αυτού και τότε η Κομισιόν ήθελε μια απορρίθμιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ο Υπουργό είπε τότε πω η προστασία των πολιτών, η προστασία καταναλωτών είναι κάτι σημαντικό, επίση σημαντικό. Και η επιχειρηματολογία την οποία προβάλλατε σήμερα, δηλαδή πω αν έχουμε πολλές διαφημίσει, τότε ο πολίτης μπορεί να βρει κάποιον άλλο σταθμό. Πιστεύω ότι πάσχει λίγο το επιχείρημα αυτό. Και πρέπει να μιλήσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό και κυρίως το επιχείρημά σας πως θα χρειαζόμασταν περισσότερη ευελιξία επειδή από άλλα κράτη έχονται άλλοι κανόνες, δηλαδή από πότε. Από πότε εμπνεόμαστε από άλλα κράτη. Από πότε αφήνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας προδιαγράψουν πώς θα δημιουργήσουμε εμείς τους δικούς μας κανόνες. Θα πρόσεχα λίγο περισσότερο με τέτοιες επιχειρηματολογίες όπως τη δική σας. Περισσότερη ευελιξία δεν σημαίνει κατά ανάγκη περισσότερα δικαιώματα καταναλωτών, αλλά περισσότερα δικαιώματα για τους επιχειρηματίες. Και σε αυτούς τους νέους τομείς βλέπουμε, όταν βλέπουμε παραδείγματο χάρη τη συγκέντρωση στοιχείων, δεδομένων, μέσω διαφήμιση, μέσω νέων δυνατοτήτων. Εκεί πιστεύω αυτό πρέπει να ληφθεί επίση υπόψη και πρέπει να διερωτηθούμε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό. Επί του παρόντος συζητούμε επίσης την οδηγία για τα ψηφιακά περιεχόμενα και αυτοί είναι τομείς οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Τι συμβαίνει με αυτές τις online υπηρεσίες λήψης δεδομένων που λένε ότι δεν χρειάζεται να πληρώσετε επειδή εμεί χρηματοδοτούμαστε από τη διαφήμιση. Αν δεν θέλετε διαφήμιση τότε πρέπει να δηλωθείτε. Και εκεί έχουμε πάλι αφαίρεση δεδομένων, συγκέντρωση δεδομένων. Είναι ερωτήματα που έχουν σημασία, την οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε εδώ. Και έχω την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επιχειρηματολογία της παραδιευκολύνει τον εαυτό της. Και πιστεύω πως θα κοιτάξουμε με μεγάλη ακρίβεια τα ερωτήματα αυτά, κάτι ακόμα, και μετά θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι. Σας κατάλαβα σωστά. Η προστασία ανηλίκων είναι καλύτερο να γίνει μεταξύ κωδίκων δεοντολογίας και όχι μεταξύ μεσορύθμιση. Δεν είμαι σίγουρη ότι σας κατάλαβα σωστά, αλλά εκεί θα έβαζα ένα τεράστιο ερωτηματικό. Καία Κάλλα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θέλω να ρωτήσω για την προστασία των ανηλίκων. Ο πάροχος της πλατφόρμας θα πάρει, θα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, αλλά λέει υπό την αίρεση της οδηγίας. Πώς είναι δυνατόν αυτό να ευθυγραμμίζεται με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να λέει ότι δεν υπάρχουν ε, υποχρεώσεις ελέγχου. Τι εννοεί η Κομισιόν. Αν δεν υπάρχει συνεχής έλεγχος ολόκληρου του περιεχομένου, πώς θα επιτευχθεί αυτή η προστασία και η ελευθερία στην ενημέρωση και στην έκφραση. Αν δεν υπάρχει ευθύνη editorial. Αντί λοιπόν για τη γενική υποχρέωση, ίσως θα ήταν προτιμότερο να λέμε ότι για τα βίντεο θα πρέπει να υπάρχει μια ειδοποίηση ότι δεν είναι κατάλληλα για τους ανηλίκους και να προσφέρονται επιλογές ε, γονικής άδειας. Ο κύριος ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση από κοντά και στενά. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, έχω μια ερώτηση. Από πλευρά της Δανίας, είναι υποαμφισβήτηση αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καλή εμπειρία Υπάρχει κάποια αξιολόγηση, κάποια εκτίμηση, κάποια εμπειρία έχετε για το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Στη Δανία τουλάχιστον έχουμε ένα εθελοντικό σύστημα συνεργασίας με τους παραγωγούς, με τους παρόχους Οπότε η ερώτηση μου είναι, γιατί να υπάρχει αυτή η αρχή της ρήτρα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση των διαφορετικών προτάσεων στην Επιτροπή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να μην υπάρξει λανθασμένη εντύπωση θέλω να πω για το ΕΛΚΑ ότι εμείς ε, σε σχέση με την προσέγγιση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο για την οδηγία για τα οπτικοακουστικά, αλλά και για τα άλλα στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν πιο πριν, συμφωνούμε επί της αρχής. Ε. Μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο πρέπει αυτά να συνεξεταστούν. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την οδηγία για τα οπτικοακουστικά διότι είναι αδιαμφισβήτητο, έχουμε μια μεγάλη συγχώνευση γραμμικών και μη γραμμικών προσφορών υπηρεσιών ενώπιόν μας. Και αν δούμε τα πράγματα με αυτό το σκηνικό προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι ένα τομέα τον έχουμε αφήσει αρρύθμιστο, και τον άλλον τον έχουμε ρυθμίσει σε ε, επαρκώς και η συνέπεια πρέπει να είναι ότι πρέπει να πορευτούμε με τη μέση, μέσω της μέσης οδού ώστε να μπορέσουμε αυτά τα περιεχόμενα εκπομπών να τα καλύψουμε ισο, ισοδύναμα αναλογικά και γι' αυτό λοιπόν είναι θετική αυτή η προσέγγιση. Δεύτερο στοιχείο που είναι σημαντικό για μας, μεγάλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γλώσσα τους, με την ισχύ τους στο πολιτισμικό, πολιτιστικό τομέα, ακόμα και και χωρίς ε, ε, προστασία στον τομέα των οπτικοακουστικών στο μέλλον χωρίς κανένα πρόβλημα θα μπορούν να παρέχουν τα προϊόντα τους σε ταινίε και μουσικά προϊόντα. Για μικρότερα κράτη θα είναι δυσχερέστερο το εγχείρημα. Αυτή η τροποποίηση λοιπόν της οδηγίας δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι οι μικρότεροι ε, πολιτισμοί, οι μικρότερα, μικρότερες εμβέλειας προϊόντα θα πρέπει να υφίστανται αρνητική διακριτική μεταχείριση. Πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε τι πρέπει να γίνει σε σχέση με μικρότερες προσφορές ε, να παραμείνουν στην αγορά και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Υποθέτω ότι για αυτόν τον λόγο έχει προτείνει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ίσως θα μπορούσε να αναφερθεί σε αυτό το θέμα ξεχωριστά η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Ροζιέρ. Νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που προσπαθούμε να πλησιάσουμε στις συνθήκες ε, για τη γραμμική και μη γραμμική μετάδοση. Αλλά θέλω να επανέλθω στις πλατφόρμες, σε αυτόν τον όρο. Που είναι διανομής οπτικοακουστικού υλικού χωρίς όμως να επομίζονται καμία ευθύνη. Λέμε ότι είναι τεχνικοί φορείς, είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν το περιεχόμενο, το τοποθετούν δηλαδή, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο την τοποθέτησή του. Ναι, αλλά τελικά βλέπουμε ότι δεν έχουμε την επιμέλεια που χρειάζεται προκειμένου να αφαιρέσουμε ε, είτε πρόκειται για περιεχόμενο παράνομο, είτε πρόκειται για σεξιστικές ε, παρεμβάσεις ή περιστρομοκρατίες, οτιδήποτε. Είναι διαφορετικά τα θέματα, αλλά δεν έχουμε την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε. Γιατί δεν υπάρχει ευθύνη. Δεν είναι οι εκδότες, ποιοι έχουν την ευθύνη. Αυτοί οι φορείς τελικά καθορίζουν κριτήρια δικά τους, που δεν έχουν καμία σχέση με τον νόμο θεωρούν ότι κάποια περιεχόμενα μπορεί να σοκάρουν, για παράδειγμα, οπότε αποφασίζουν να αφαιρέσουν κάποιο περιεχόμενο hm. τότε ας πούμε που είχε εξαφανιστεί ο πίνακας που αναφερόταν στην καταγωγή του κόσμου. Δεν είναι όμως κάτι που ήταν κατά του νόμου, οπότε πρόκειται για λογοκρισία ή που έχουμε λογοκρισία, αν πρόκειται από τους ε, τεχνικούς που αφαιρούν ε, περιεχόμενο ή αλλιώς πρόκειται για πραγματικούς εκδότες. Γι' αυτό λοιπόν θέτω το θέμα αυτό της πλατφόρμας, γιατί έτσι καταλήγουμε σε ανόητες και παράλογες καταστάσεις, δεδομένου ότι κανείς τελικά δεν έχει την πραγματική ευθύνη. Πρόεδρος, θέλω και εγώ να ρωτήσω μερικά πράγματα. Χαίρομαι που βλέπω το άρθρο 6α και 28α, που αναφέρονται στην προστασία των ανελίκων από το περιεχόμενο. Περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για ανελίκες, για τις πλατφόρμες, video sharing κλπ. Στο πακέτο τηλεπικοινωνιών είχαμε μιλήσει πάρα πολύ για το θέμα της γονικής άδειας και πολλοί έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να δίνεται αυτό στους γονείς γιατί μπορεί να καταλήξει στον αποκλεισμό κάποιου περιεχομένου. Εγώ νομίζω ότι οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται και αν θέλουν να επιβάλλουν αυτούς τους ελάχους. Μπορείτε λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε ότι εδώ δεν θα κάνουμε κάτι αντίθετο από αυτό που είχε συμφωνηθεί στο δέσμι για τις τηλεπικοινωνίες και θα εξασφαλίσουμε ότι οι γονείς μπορούν να προστατεύσουν τους ε, ανήλικες για την αρχή της χώρας προέλευσης. Οι πάροχοι υπηρεσιών λένε ότι φορολογούνται ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Γιατί το προτείνετε αυτό. Και αυτό το 12% 12 λεπτά ανά ώρα υπολογίζεται σε 24 ώρες βάση, δηλαδή μπορείς ε, μία μόνο στιγμή της ημέρας να έχεις όλες σου τις διαφημίσεις και να καταλήξεις να έχεις μια ώρα συνεχώς διαφημίσεις και τίποτα άλλο. Δεν είναι αυτό που θέλουμε φαντάζομαι. Από την Επιτροπή τώρα θέλετε να μας παρουσιάσετε τις πλατφόρμες. Δεν κατάλαβα ότι... Σας το είχαμε ζητήσει, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι θα το κάνετε. Μια στιγμή. Για απαντήστε πρώτα κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις παρακαλώ για το οπτικό ακουστικά και μετά θα δούμε. Λοιπόν, παρακαλώ απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα σας διευκρινίσω κάποια πράγματα που καταλαβαίνω τώρα ότι δεν ήταν ξεκάθαρα. Για την πρώτη ερώτηση, όσον αφορά το θέμα της ε, διαφήμισης, λέτε ότι θέλετε απορρίθμιση στη διαφήμιση. Έχει γίνει αξιολόγηση αντικτύπου, άρα ξέρουμε τι ακριβώς προτείνουμε. Ειλικρινά δεν πιστεύουμε ότι η σημερινή κατάσταση είναι συγκρίσιμη με την κατάσταση που είχαμε πριν από πόσα χρόνια. Το 2007, με εφαρμογή το 2009. Η αγορά δεν είναι ίδια καθόλου όπως τότε. Έχουμε αναλύσει την ελαστικότητα της ζήτησης έχουμε αναλύσει την επιθυμία των ε, καταναλωτών να αποφύγουν τις διαφημίσεις, να στραφούν. Όχι, δεν λέμε βάλτε διαφημίσεις 20 λεπτά. Όχι. Λέμε κάντε μόνοι σας τη διαχείριση του χρόνου. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση γιατί η αξία της ε, διαφήμισης ανεβαίνει όσο πιο λίγο είναι ο χρόνος. Όσο πιο πολύ χρόνος υπάρχει για διαφήμιση, τόσο μειώνεται το κόστος της διαφήμισης. Οπότε λέμε ότι οι broadcasters αυτοί οι ίδιοι θα πρέπει οικονομικά να ε, αναλύσουν το θέμα και να δουν τι τους συμφέρει. Τώρα, αν σε μια χώρα μέλος, κάποια χώρα μέλος θεωρεί ότι η εξέλιξη της αγοράς τους δεν είναι σε αυτό το στάδιο, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση, μπορούν να κρατήσουν τους δικούς τους κανόνες. Όσον αφορά τώρα το product placement, την ε, κρίζα διαφήμιση, Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Α, μάλλον όχι, γι' αυτό το επιχείρημα. Λέτε ότι αν υπάρχει περισσότερη γκρίζα διαφήμιση από τι ΗΠΑ και εμεί πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Δεν είπα αυτό. Και σίγουρα δεν εννοούσα αυτό. Αυτό που λέω είναι ότι η γκρίζα διαφήμιση σήμερα τι κανόνε έχει. Λένε, απ' τη μια, ότι δεν θα πρέπει να γίνεται τέτοια έτσι κυρίαρχη γκρίζα διαφήμιση και λέει ότι αν έχετε τέτοια κρίση διαφήμιση πρέπει και τον προτέρων να ενημερώνετε τον καταναλωτή, το θεατή. Αν έχετε λοιπόν μια ευρωπαϊκή παραγωγή, μπορείτε πού θα διαφημίσετε το προϊόν σας με αυτή την κρίση διαφήμιση και μπορείτε να το ανακοινώσετε πριν. Όταν όμως κάτι έρχεται απ' έξω από οποιαδήποτε χώρα, δεν έχει σημασία, για να παρέμβετε στο επίπεδο της παραγωγής αυτό είναι πιο περίπλοκο. Γι' αυτό και καταλήξαμε στην εκτίμηση που κάναμε ότι οι κανόνες εφαρμόζονται από τους ρυθμιστές με διαφορετικούς τρόπους. Γιατί τι σημαίνει κυρίαρχη γκρίζα διαφήμιση. Με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό αυτό που λέμε τώρα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα στην αγορά, ότι υπάρχει γκρίζα διαφήμιση και ότι είναι πιο εύκολο να επιμείνουμε στη διαφάνεια. Δηλαδή, ενημερώστε το θεατή σας ότι υπάρχει τέτοια γκρίζα διαφήμιση. Αυτό. Διευκρινήσει τώρα για την προστασία των ανηλίκων. Είπα ότι πρέπει να γίνεται αυτό μέσω κωδικών και ναι και όχι. Όχι γιατί οι κανόνες για την προστασία των ανηλίκων για τις ε, γραμμικές υπηρεσίες είναι κάτι για το οποίο υπάρχει ζήτηση. Δεν πρέπει να μπορούν να δουν κάποιο περιεχόμενο οι ανήλικοι και αυτό υπάρχει σαν ρύθμιση. Τώρα προσθέσαμε το άρθρο 6 που είναι κάτι νέο που λέει ότι ενθαρρύνουμε να εφαρμόζεται η ρύθμιση. Το νέο άρθρο επίσης λέει ότι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για την βλάβη που μπορεί να πάθει ο Μανίλικος αν δει κάποια συγκεκριμένη ταινία που έχει βία, σεξ, ναρκωτικά, δεν ξέρω εγώ τι. Θα υπάρχει η πληροφορία αυτή. Οπότε οι γονείς να μπορούν ανάλογα να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν ή όχι. Αυτό λοιπόν ενθαρρύνουμε να υπάρχει. Το θέλουμε στη ρύθμιση. Αυτό εννοούσα επιστρέφω στις ερωτήσεις για την προσβασιμότητα. Όσον αφορά το gap. Η σημερινή, το κενό μάλλον ανάμεσα στον ένα κανονισμό και στον άλλο, στη μία ρύθμιση και στην άλλη. Όσο δεν υπάρχει νέο νομικό μέσο, ισχύει το παλιό. Καταλάβαμε ότι υπάρχουν κάποιοι φορείς που θέλουν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση για τα οπτικοακουστικά. Η Κομισιόν είπε ότι θέλει να τα βάλει χωριστά. Αν ο νομοθέτης αποφασίσει κάτι άλλο, τότε θα συμπεριληφθούν και τα οπτικοακουστικά. Για τις πλατφόρμες. Τι σημαίνει video sharing platform. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί όπως έλεγα δεν πρόκειται για όλες τις πλατφόρμες. Εμείς θεωρούμε ότι τα οπτικοακουστικά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Η εικόνα είναι κάτι πολύ δυνατό. Γι' αυτό και έχουμε μια ειδική οδηγία για αυτούς ακριβώς τους τομείς. Και πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο και στον κόσμο online. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό οι πλατφόρμες αυτές που είναι η αναμετάδοση οπτικοκουστικού υλικού με σκοπό το, κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση. Οπότε άλλο είναι οι πλατφόρμες ιδιωτικού τύπου μεταξύ φύλων. Και κάτι άλλο σημαντικό, αν δεν υπάρχει ευθύνη περιεχομένου, μπορούμε να προσθέσουμε κάτι το οποίο να λέει ότι ο πάροχος έχει κάποιον έλεγχο της παρουσίασης και του ελέγχου αυτού που προσφέρει. Αυτό κάνει τη διαφορά με μια απλή φιλοξενία, θα έλεγα, που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Τώρα, οι ώρες πώς μετρούνται. Δεν το έχουμε καθορίσει αυτό ακόμα. Μέχρι τώρα πώς λειτουργεί. Κάποιες χώρες μέλη έχουν ήδη, αρκετές μάλιστα, 16, ήδη βάζουν ώρες, μετράνε, με διαφορετικούς τρόπους. Άλλες με κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο είναι, υπολογίζεται χωριστά. Άλλοι υπολογίζουν το χρόνο που κρατάει ε, το κάθε επεισόδιο. Δεν επιβάλλεται κανένα σύστημα ακόμα γιατί το άρθρο 13 δεν επιβάλλει κάποιο σύστημα. Άρα μένει να το δούμε ακόμα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα συστήματα στις διάφορες χώρες αλλάζουν. Πάντως, ή ανά επεισόδιο, ε, με το χρόνος, ή ανά χρόνο. Αυτές οι δύο επιλογές υπάρχουν προς το παρόν για τη μέτρηση των ορών. Τι άλλο, ναι. Υπάρχει επίσης... Α, ναι, να διευκρινίσω και κάτι. Για το 20%. Είναι μόνο για τη μεζήτηση υπηρεσίες, δεν είναι για τις video sharing platforms. Τώρα, πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε βάση προβλήματος. Εντοπίζουμε πρόβλημα και μετά δρούμε. Δεν νομοθετούμε έτσι γενικά εν κενό. Όταν εντοπίζουμε κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα την προστασία των ελίκων, δρούμε. Για την διαφήμιση σήμερα ήδη υπάρχει ένα νομικό μέσο που είναι η οδηγία για τις εμπορικές πρακτικές. Και εντοπίσαμε ότι κάποιες χώρες μέλη, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ήδη τα έφερε κατευθυντήρες γραμμές η Επιτροπή, πώς να εφαρμοστεί στον online κόσμο. Άρα έχει γίνει η αρχή. Πώς να εφαρμοστούν οι κανόνες για την προστασία των παιδιών στις υπηρεσίες on demand. Το μόνο μέτρο δεν είναι να πούμε ότι πριν από κάποια ώρα, για παράδειγμα, δεν θα μπορούν να δουν. Τα κείμενα λένε ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Και έχετε δίκιο που λέτε ότι σε πολλές χώρες συζητιούνται τα μέτρα με τον κλάδο. Στις κατοχώρες, για παράδειγμα. Ολοκληρώστε παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, μετά. Για να δούμε τώρα για τη λογική των ε, ποσοστώσεων. Δεν πιστεύουμε ότι στον demand οι ποσοστώσεις είναι το τέλειο. Γιατί μπορείς να έχεις το 80% μαζεμένο. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να προβάλλουμε το περιεχόμενο. Αν δεν έχει ούτε ένα μίνιμουμ, τότε πώς θα το θεωρήσεις κυρίαρχο. Βάζουμε λοιπόν το 20% σαν μια υποχρέωση. Υπήρχε και μια πολύ καλή ερώτηση που κάνατε για το ότι οι πλατφόρμες σήμερα δημιουργούνται βάσει των ε, ιδίων τους κριτηρίων για το τι είναι ε, βλαβερό και τι όχι ως περιεχόμενο. Εμείς εφαρμόζουμε τόσο αναφέρει η οδηγία, για παράδειγμα για την υποκίνηση στο μίσος. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα, δεν αφαίρετο. Με ρωτήσατε για το χώρο προορισμού. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι σχετικό με τη μεταφορά στη χώρα προορισμού. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι κάποιες διατάξεις που θυμίζουν ε, πολύ φορολογικά πρέπει να ακολουθούν την ίδια αρχή. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα μας. Εξού και περιοριστήκαμε μόνο σε αυτήν τη διάταξη που έχει να κάνει με την εισφορά. Πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την λεπτομερή παρουσίαση. Μια πρόταση διαβιβάστε τη στην Επιτροπή. Όταν έρχεστε να παρουσιάσετε προτάσεις από την Επιτροπή σε εμά, είναι επικοδομητικό να υπάρχει μια σειρά σημείων με bullet points με τα πιο σημαντικά από όσα έχετε να παρουσιάσετε αυτό το θέμα μεταξύ της ε, AVMS και των πλατφορμών ε, ε, της ομάδας δηλαδή θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο παρουσίασης και τώρα λίγη ο χρόνος πλέον γιατί έχει προγραμματιστεί συνάντηση συντονιστών και δεν έχουμε τώρα τον χρόνο για την παρουσίαση για τις πλατφόρμες. Νομίζω ότι θα θέλαμε να συνεχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε σε άλλη συνάντηση να καλύψουμε τις πλατφόρμες και να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος. Δεν θέλω να επιστρέψει στην Επιτροπή και να δημιουργηθεί εντύπωση ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τις πλατφόρμες. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και έντονα μάλιστα, ιδιαίτερα τα θέματα τα οποία αφορούν την προστασία των καταναλωτών και της ενιαίας αγοράς και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα για τα στοιχεία της εσωτερικής ενιαίας αγοράς ε, υπό το AVMS. Νομίζω ήταν σημαντικό αυτό. Και ευχαριστώ και προσβλέπω Αδειμονώ να έχουμε αυτή την επαφή. Μια σαφή παρουσίαση από την Επιτροπή για τις πλατφόρμες την επόμενη φορά. Πρέπει να περάσουμε τώρα και κλεισμένων των θυρών στη συνάντηση των συντονιστών. Αν δεν ανήκετε στο πλαίσιο των ε, μελών αυτής της συνάντησης, παρακαλώ να αποχωρήσετε. Um,